Good afternoon, dear colleagues. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Είναι λίγο περίεργη αυτή η αίθουσα που μας δώσαν. Προσπαθώ να εντοπίσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για να ξέρω που κάθεστε. Τέλος πάντων τι να κάνουμε, αυτοί μας δώσαν. Να ξεκινήσω με την έγκριση της σημερινής σας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, την εγκρίνουμε. Διερμηνία υπάρχει προς 16 γλώσσες και η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή με το συνήθι τρόπο. Να κάνω τις εξής ανακοινώσεις και σε σχέση με τη συνάντηση των συναντιστών που έγινε σήμερα το πρωί. Θα διοργανωθεί νέα ακρόαση 16 ε, Ιουνίου, η κυρία Ντόρο Τεσάρ, η κυρία Σαμπίντο και ο Όλιβερ ε, Χομπίντο, ο Πόρχης Καϊ από το Πανεπιστήμιο Ασάφ, του Ασάφενμπουργκ και ως συνήθως θα αποσταλούν γραπτές ερωτήσεις στους προσκεκλημένους και θα σας αποσταλούν πριν από τη συνεδρίαση. Να σας πω επίσης ότι με βάση τη συζήτηση που είχαμε το πρωί θα ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε όλοι οι εμπειρογνώμονες και μάρτυρες που ε, έρχονται ε, θα συμμετάσχουν στην, στις ακροάσεις μας. Ήρθα σε επαφή και με τον πρόεδρο της Επιτροπής ΙΜΚΟ για να συντονιστούμε καλύτερα όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το πλαίσιο έγκρισης τύπου. Οι, ερωτές, οι ερωτήσεις, ε, το ερωτηματολόγιο λοιπόν θα αποσταλεί στην αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο και συντάσσουμε σε συνεργασία με τους συντονιστές και τον εισηγητή. Θα σταλεί και στο Κοινό Κέντρο Έρευνας ένα αίτημα γιατί θεωρούμε ότι οι πληροφορίες που μας δόθηκαν από την υπηρεσία αυτή δεν είναι επαρκής. Ενώ όλη η αλληλογραφία της Επιτροπής ΕΜΙΣ θα δημοσιεύεται από εδώ και στο εξής στο διαδίκτυο. Έχετε σχόλια? τα πρακτικά της συνεδρίασης της 19ης Απριλίου βρίσκονται στο διαδίκτυο. Αν δεν υπάρχουν σχόλια θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται και αυτά. Οπότε μπορούμε να περάσουμε και στο πρώτο τμήμα της σημερινή ακρόασης και θα ήθελα θερμότατα να ε, καλωσορίσω τον κύριο Ρίτσαρτ Σμόκερς, σύμβουλο, και τον ε, κύριο Ρομπ Κουλενάρε, της Ολλανδικής Οργάνωσης Εφαρμοσμένης Επιστημονικής Έρευνας, TNO. Όπως πάντοτε, έχουμε στη διάθεσή μας μία ώρα και 15 λεπτά και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Ρίτσαρτ Σμόκερς για 10 λεπτά και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με την ακρόασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρόσκληση που μας απίφθηνε. Θα σας ε, παρουσιάσω, θα σας κάνω μια παρουσίαση. Δεν θα ε, μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες όσον αφορά τη, τη, τα στοιχεία που εμφανίζονται στις διαφάνειες για να αφήσω χρόνο για τη συζήτηση. Να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα των μετρήσεων που κάναμε για τις ε, εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου, των διζελοκινητών, των ε, αυτοκινήτων τόσο ε, σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές. Είμαστε ανεξάρτητος ε, ερευνητικός οργανισμός με 3.000 εργαζόμενους μεταξύ αυτών των τομέων που μας απασχολούν είναι και οι μεταφορές και το logistics όπου και προβαίνουμε σε διάφορες ε, αξιολογήσεις που σχετίζονται με τις, μεταβο... με τις ε, οδικές μεταφορές. Μια σύνοψη. Να δείτε εδώ ότι έχουμε μετρήσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι και επιβατικά και εμπορικά, εμπορικής χρήσης αυτοκίνητα, σε, ε, σε πραγματικές συνθήκες και σε συνθήκες εργαστηρίου. Οι εκπομπές που μετρήσαμε είναι πολύ ψηλότερες από αυτές που προκύπτουν από τις ε, δοκιμές έγκρισης τύπου ε, κατά τρεις έως τέσσερις φορές σε ορισμένε περιπτώσεις. Για το ε, Euro 6 είναι 2 έως 6 φορές και κατά 6 φορές για το, για το Euro 5 κατασκευής 2010-2011, κατηγορία 1 και 2 εξετάσαμε διάφορες μάρκες αυτοκινήτων και διάφορα μοντέλα. Το πρόγραμμά μας το εκπονήσαμε για το Ολλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε εμπειρία 30 χρόνων και έχουμε εξετάσει μια σειρά από ε, παράγοντες ρήπανσης, ε, φορτηγά, ελεοφορία ε, εμάς στόχος μας, κύριος στόχος μας είναι να εξετάσουμε και να μετρήσουμε τις ε, εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να τροφοδοτούμε τα στοιχεία αυτά ε, για διάφορες μελέτες για την χάραξη πολιτικής δημόσιων φορέων της, των κάτω χωρών. Επίσης, εξετάζουμε νέες τεχνολογίες, για παράδειγμα μετρήσεις ε, διέγερσης και συμμετέχουμε και στην ε, εκπόνηση νέων κανονισμών στις ε, Βρυξέλλες. Επίσης, εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και μια φωτογραφία από το 1970, όταν ξεκινήσαμε αυτές τις δοκιμές. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι πολύ πιο ε, σύγχρονα. Έχουμε δικές μας ε, μετρήσεις, χρησιμοποιούμε PEMS και το 2014 δημιουργήσαμε και μια απλοποιημένη μέθοδο μέτρησης ε, σε πραγματικές συνθήκες με τίτλο SEMS για τη μέτρηση των εκπομπών των οχημάτων. Αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει υπάρξει ε, μια εξέλιξη των οχημάτων τα οχήματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, το ίδιο βεβαίως ε, ισχύει και για τις ε, μεθόδους μετρήσεων. Και αυτό που χρειάζεται να πούμε είναι ότι οι μετρήσεις στο δρόμο ε, κατέστησαν δυνατές το 2011 μόλις, όταν και αποκτήσαμε τον εξοπλισμό PEMS. If you look at vehicle όπως είπα, τα οχήματα έχουν γίνει πολύ περίπλοκες, πολύ προπλοκά μηχανήματα με ηλεκτρονικά κυκλώματα, δεν είναι πλέον απλά ένα μηχάνημα με έναν απλό ε, κινητήρα και γι' αυτό το λόγο είναι και πολύ πιο περίπλοκη η μέθοδος για τη μέτρηση των οξυδίων του ε, αζότου. Τα πρότυπα PM που συζητούνται και εδώ σε αυτή την Επιτροπή ε, είναι εκείνα που οδήγησαν στην ε, διασπορά και την ευρύτατη χρήση των PM, ε, κάτι που οδήγησε σε πολύ χαμηλές εκπομπές σε σύγκριση με τα πετρελοκίνητα οχήματα του Euro 5, αλλά για, τα, για τις εκπομπές αζότου, οξυδίων του αζότου, τα, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Βασικά όλα τα οχήματα που ε, ε, μετρήσαμε παρουσίασαν αυξημένα σε εκπομπές οξυδίων του αζότου, όχι απλά σε ποσοστιαία βάση, αλλά κατα ε, κατά 2-3 έως και έξι φορές. Επίσης, μια συνήθιση συμπεριφορά είναι αυτή, αν χρησιμοποιεί κανείς Έχουμε διαπιστώσει ότι σε έναρξη θερμής ε, ε, εκκίνησης μιας, ε, ενός κινητήρα οι εκπομπές είναι υψηλότερες από ότι στην αντίθετη περίπτωση. χάρη στα ΠΕΜΣ ε, ε, ε, δεν χρειάζεται πια να, κάνουμε ε, τις μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες. Στο δρόμο δηλαδή. Euro 6. Αυτό που βλέπουμε είναι μια τι εικόνα. Κάποια οχήματα είναι καθαρά, κάποια άλλα εξαρτώνται από τον κύκλο οδήγησης, αλλά γενικά παρουσιάζουν μια σταθερή εικόνα ως προς τις εκπομπές τους ε, πάνω από το όριο βέβαια, με μία και μόνο ε, εξαίρεση. Γενικά η, η εικόνα είναι ε, σταθερή, ομοιόμορφη για όλα τα οχήματα που ε, ελέγξαμε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για το ζήτημα που μας απασχολεί. Εδώ βλέπετε τις εξελίξεις των, των εκπομπών NOx το όριο για τα, για τα τζελοκίνητα ήταν υψηλότερο από ό,τι για τα πετρελαιοκίνητα. Άμα δείτε εδώ στην ε, πράσινη ράβδο, βλέπετε τις ε, εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου που είναι σταθερά χαμηλότερες από το, όριο που, το επιτρεπόμενο όριο και άμα δείτε την, ε, την μπλε ράβδο, αυτά είναι τα τζελοκίνητα αυτοκίνητα, κάτω από το όριο για το Euro 1 και Euro 2, αλλά πάνω από το όριο για τα Euro 3 έως Euro 6. Και άμα δείτε από το Euro 1 ε, ε, έως το Euro 5, το όριο έχει μειωθεί κατά 5 φορές, ενώ οι εκπομπές έχουν μειωθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό. Το Euro, το Euro 6, η εικόνα που παρουσιάζει είναι κάπως καλύτερη, αλλά ε, η τάση παραμένει η ίδια. Οι εκπομπές ε, είναι πολύ υψηλότερε όταν εξετάζονται, όταν, δοκι... όταν, μετρώνται, ε, όταν μετρώνται σε πραγματικές συνθήκες στο δρόμο. Η εικόνα που προκύπτει για εμάς από αυτά που έχουμε δει είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι κατασκευαστές βελτιστοποιούν το hardware και το software των ε, οχημάτων με βάση την διαδικασία μέτρησης των δοκιμών αφορά το φορτίο του κινητήρα και αυτό δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιείται το hardware και το software του κινητήρα ε, και έτσι τα αυτοκίνητα αυτά φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα στις δοκιμές αλλά όχι στις πραγματικές συνθήκες. Εμείς δεν έχουμε δει ε, συσκευές αναστολής. Ε, δεν, μπορούμε, δεν έχουμε σαφείς ενδείξεις τουλάχιστον. Πάντως γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι εκπομπές είναι υψηλότερε στις πραγματικές συνθήκες από ό,τι στο εργαστήριο. Εδώ βλέπετε και ένα γράφημα. Εδώ ο οριζόντιος άξονας δείχνει το πλάτος, το εύρος μάλλον των ε, φυσιολογικών συνθήκων οδήγησης. Ε, αυτές δηλαδή που προκύπτουν ε, σε πραγματικέ συνθήκε στον δρόμο και ε, οι προποθέσει τύπου καλύπτουν μόνο ένα πολύ συγκεκριμένο ε, τμήμα αυτών των, των συνθήκων. Αυτό που βλέπουμε από τις μετρήσεις μας είναι αυτό που βλέπετε εδώ στις πράσιν, στην πράσινη και στην ε, μπλε γραμμή ότι τα πράγματα δηλαδή πάνε καλά όταν ε, οι συνθήκες προσωμιάζουν με εκείνες των δοκιμών, ενώ όταν οι συνθήκες γίνονται πιο σοβαρές, πιο αντίξωες, ε, τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι πολύ πολύ χειρότερα. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι οι εκπομπές κυμαίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και το αστείο είναι ότι οι, οι ψηλότατες αυτές εκπομπές που θα περίμενε κανείς ότι η νομοθεσία ε, θα είχε ως σκοπό το αντίθετο, δεν ρυθμίζεται καθόλου νομοθετικά πουθενά. Ένα άλλο πράγμα που, που δεν απαιτείται από τους, αυτοκιν, από τις αυτοκινητοβιομηχανίες είναι ότι δεν αποτελούν ευθύνη τους τα οχήματα αφού φύγουν από το εργοστάσιο και αυτό αφορά τη συμμόρφωση, την ε, ανθεκτικότητα κτλ. κτλ. Όταν τους ε, θέτουμε το ζήτημα αυτό, ε, μας ε, λένε ότι... όταν τους λέμε δηλαδή ότι οι εκπομπές των οχημάτων τους υπερβαίνουν αυτά που ισχυρίζονται οι ίδιοι, λένε ότι οι ίδιοι συμμορφώνονται με, την, με τις δοκιμές που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ποιες είναι οι επιπτώσεις όλων αυτών. Οι επιπτώσεις των υψηλών εκπομπών είναι ότι οι πόλεις δεν έχουν καταφέρει να επιτύχουν τους στόχους για, την, ε, ε, για, την, ε, για τον καθαρό αέρα. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται υψηλές συγκεντρώσεις οξυδίων του αζότου μέσα στις πόλεις. Ταυτόχρονα όμως ε, μειώνεται η αποτελεσματικότητα διαφόρων μέτρων πολιτικής που μπορούν να χαράξουν και να εκπονήσουν οι πόλεις προκειμένου να ε, αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά προβλήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ε, ένα, μια πολύ μεγάλη λύση, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. πρόκειται η λύση αυτή θα είναι και χρονοβόρα και δαπανηρή. Και αυτό πρέπει να τονιστεί, γιατί νομίζουμε ότι δεν έχει τονιστεί επαρκώς τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ολλανδίας έχουμε ζητήσει αναθεώρηση όλων των ε, ε, μετρήσεων δοκιμής που γίνονται τα τελευταία χρόνια, από το Euro 4 δηλαδή, το έχουμε κάνει αυτό στην Ολλανδία, βλέποντας, ε, δείχνοντας τα αποτελέσματα ε, σε διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Έχουμε παρουσιάσει τα πορίσματα των ερευνών μας σε ομάδες εργασίες. σε φορείς χάραξης πολιτικής. Ε, έχουμε ενημερώσει το Κοινό Κέντρο Έρευνας για όλα αυτά και άλλα ερευνητικά κέντρα που, που ασχολούνται με τις εκπομπές. Έχουμε διοργανώσει και κάποιες διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους φορείς και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως έχουμε παρουσιάσει τα ευρήματά μας και στον τύπο. Τελευταία διαφάνεια, τελευταίο ερώτημα βεβαίως είναι. Ποιες είναι οι εξελέξεις σε σχέση με την ομοθεσία από εδώ και πέρα και αν θα βοηθήσουν. από την εμπειρία μας, ε, ακόμα και οι νέες μέθοδοι μέτρησης που προτείνονται εξακολουθούν να είναι εργαστηριακές και από αυτή την άποψη δεν μπορούν να λύσουν πλήρως το περιβαλλοντικό πρόβλημα, γιατί πάλι θα υπάρχει τρόπος να βελτιστοποιείται. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι ε, πρόκειται για μια καλή αρχή, ξεχωριστή ε, αξιολόγηση των των, ε, των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες είναι απαραίτητη και κάτι που έχει χαθεί λίγο στη συζήτηση είναι ότι δεν θα πρέπει να ε, ελέγχεται μόνο η συμμόρφωση αλλά θα πρέπει να ε, αναθεωρηθούν και να ξαναελεγχθούν οι, όλες οι μέθοδοι μετρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των εκπομπών. Από αυτή την άποψη, ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός είναι σημαντικός. Αυτά ήθελα να πω. Thank you very much. It's been a few minutes more. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα εισήγηση. Να ακούσουμε τώρα τους εισηγητές. Ο κύριος Σάλμπα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σμόκερς. Είναι προφανές ότι οι δικές σας... Α, περιμένατε λίγο. Εντάξει, ακούτε τώρα. Ωραία, μπορείτε να συνεχίσετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριε Σμόκε. Ευχαριστώ πολύ ε, για την εισήγησή σας ε, που μας ενημερώσατε για τις διαρκείς βελτιώσεις από το ΕΡΟΕΝΑ μέχρι το Euro ε, θα γνωρίζετε βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πόσο ελλειπής είναι, ε, ελλειπές είναι μάλλον το καθεστώς αυτό ε, που ισχύει και ξεκίνησε να εξετάζει τις πραγματικές εκπομπές η Ευρώπη θα πρέπει να μετατραπεί στην πρώτη περιοχή του κόσμου όπου χρησιμοποιούνται αποδείξεις και στοιχεία σε πραγματικές συνθήκες. Ερώτηση τώρα σε σχέση με τις γραπτές ε, απαντήσεις που μας δώσατε, όπου λέτε ότι σε υψηλές ταχύτητες μπορεί να εκπέμπονται 10 με 20 φορές περισσότερο μονοξίδιο του αζότου, που είναι το όριο που ε, επιτρέπεται. Όταν μιλάτε για υψηλή ταχύτητα, ε, σε ποια ταχύτητα αναφέρεστε. Επιπλέον, θα ήθελα να ρωτήσω για μια άλλη απάντηση που δώσατε γραπτό. λέτε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι σαφή σε σχέση με τον ορισμό των ε, προβλέψουν για την απενεργοποίηση. Σε προηγούμενες ακροάσεις ε, άλλοι ειδικοί μας είπαν ότι αυτές ε, οι μηχανισμοί για απενεργοποίηση δεν μπορούν να εντοπιστούν. Άρα λοιπόν η ερώτησή μου είναι τι μπορεί να γίνει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί αν ο ορισμός δεν είναι σαφής ε, και άρα αυτοί οι μηχανισμοί δεν μπορούν να ανοιχνευτούν έχουμε πρόβλημα. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η μία σας ερώτηση αφορά τις υψηλές εκπομπές σε υψηλές ταχύτητες. Ναι, όντως ε, με τα σημερινά αυτοκίνητα όταν αυτά τρέχουν σε μεγάλες ταχύτητες στους αυτοκινητοδρόμους, δηλαδή πάνω από 130 χιλιόμετρα την ώρα, Δοκιμάζουμε δηλαδή τα αυτοκίνητα στους αυτοκινητοδρόμους ε, στη Γερμανία όπου τα οδηγούμε σε 150 χιλιόμετρα την ώρα και έτσι βλέπουμε ότι είναι πολύ υψηλότερε οι εκπομπές από ότι το ανώτατο όριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες οι εκπομπές και σας λέω ότι αυτές είναι μετρήσεις στα υπάρχοντα αυτοκίνητα. Και έπειτα πρόκειται και εκπομπές ανά χιλιόμετρο, ενώ στις αστικές περιοχές, στην αστική οδήγηση με πολλά σταμάτα ξεκίνα, έχουμε άπειρες εκπομπές ανά χιλιόμετρο. Βλέπουμε εκπομπές στις πόλεις εκεί και που τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα, ακίνητα. Τώρα, και τους ε, συσκευές αυτές και την ανείχνευσή τους, δεν ξέρω από νομικής άποψης πώς θα μπορούσε να γίνει. Για μας ε, η νομοθεσία λέει δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αυτές οι συσκευές, αλλά δεν ορίζονται, ούτε λέει πώς θα πρέπει να δοκιμάζονται και να ελέγχονται. Δεν διευκρινίζεται καμία διαδικασία για έλεγχο για την παρουσία τέτοιων συσκευών και έτσι καθίσατε δύσκολο για οποιονδήποτε να το ερευνήσει και να ισχυριστεί ότι ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί τέτοιους μηχανισμούς και να στοιχειοθετήσει ε, κατηγορία και αποδείξεις. Εφόσον δεν ορίζετε σαφώς τι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, δεν ξέρετε επίσης πώς θα το αποδείξετε. Και αυτό το πρόγραμμα που εμείς ε, τρέχουμε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει στόχο να δει ποιες είναι οι πραγματικές εκπομπές και άρα δεν θέλουμε να ερευνήσουμε συγκεκριμένα μοντέλα για να ψάξουμε τις τεχνικές οικούς λόγους για αυτά που βλέπουμε. Βλέπουμε διάφορα αυτοκίνητα για να έχουμε ε, στοιχεία για τις εκπομπές ε, για λόγους ποιότητας ε, του αέρα. Ακόμα λοιπόν και αν βρίσκαμε τους συσκευές ε, δεν θα τις ελέγχαμε γιατί είναι άλλος ο στόχος μας. Κύριε Σάλμπα, πολύ σύντομα. Επανέρχομαι στο πρώτο μου σχόλιο. Δηλαδή μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να συμφωνήσουμε πως η Ευρώπη θα είναι η πρώτη περιοχή στον κόσμο που θα χρησιμοποιεί πραγματικές, δοκιμές σε, σε πραγματικές συνθήκες. Ναι, νομίζω πως είμαστε οι πρώτοι αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει ότι πιστεύουμε πως η λύση του προβλήματος βρίσκεται στις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εφαρμοστεί με τον σωστό τρόπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, τεχνικές τεχνικές και κατάλαβα από τις απαντήσεις που μας δώσατε γραπτός και καταλαβαίνω ότι χάρη σε έναν συνδυασμό υφιστάμενων ε, τεχνολογιών τα οχήματα πρέπει να μπορούν να σεβαστούν τους κανόνες. Είναι τεχνικός εφικτό αυτό, ναι, ναι απάντηση να είναι σωστά και στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων διαπιστώνουμε πως όλα τα οχήματα τηρούν τα όρια. Δηλαδή οι εξοπλισμοί των αυτοκινήτων λειτουργούν όπως πρέπει ώστε να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο εκπομπών. Ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση και πάλι σε βάση των γραπτών σας απαντήσεων είναι αληθεύει μάλλον πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να καταργηθεί η τεχνολογία LNT και SR για να αποφύγουμε βλάβες στους κινητήρες. Ναι, μάλιστα. Δεν είναι απαραίτητο το LNT-SR να καταργηθούν, γιατί αυτά τα συστήματα λειτουργούν ανεξάρτητα από τον κινητήρα και το LNT-SR που χρησιμοποιούνται δεν έχουν αντίκτυπο στον κινητήρα. Ευχαριστώ. Τρίτη ερώτηση τεχνικής φύσης γίνεται πολλής λόγος γιατί το, τονίζεται το διοξίδιο του άνθρακα και παραμελείται το, το οξύδιο του αζότου. Είναι αλήθεια ότι επηρεάζει λιγότερο το οξύδιο του αζότου. Απάντηση, ναι. Αν βάλουμε στη ζυγαριά τα δυο, τους δύο ρήπους και δούμε το κινητήρα και πόσο αυτός θα είναι πιο αποδοτικός, Όταν χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη τεχνολογία υπάρχει αποσύνδεση, άρα στις εκπομπέ δεν υπάρχει πλέον ε, συσχετισμός ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα στο διοξίδιο και την αποτελεσματικότητα στο οξύδιο του αζότου. Τώρα αν θα υπάρχει κύρωση για το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα αν πρόκειται για τη μείωση του οξυδίου του αζότου ή του διοξιδίου του άνθρακα νομίζω ότι είναι ε, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στα στάνταρα. Θα ήθελα να επανέλθω τώρα σε κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν στην Επιτροπή. Επιτρέψτε μου να περάσω στο πολιτικό ε, επίπεδο. Διαπιστώνω στο ντοσιέ ότι από το 2010 το δική σας υπηρεσία διαπιστώνει ότι υπάρχει αύξηση των εκπομπών οξυδίου του αζότου στους δρόμους. Και παραθέτω φαίνεται πως μια άλλη στρατηγική μείωση εκπομπών του οξυδίου του αζότου θα πρέπει να εφαρμοστεί. Εσείς αυτές τις πληροφορίες τι τις κάνατε, κάνατε αυτή τη διαπίστηση, την απευθύνατε στους πολιτικούς ηθήνοντες για να τους πείτε ότι πρέπει κάτι να γίνει και αν ναι, κάναν όντω κάτι στις κατοχώρες ή στις Βρυξέλλες. Ναι, όπως σας είπα εργαζόμαστε για το ε, Ολλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όλα τα πορίσματά μας διαβιβάζονται στο Υπουργείο μας, ε, αλλά και διαβιβάζονται σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Έχουμε, ε, κάνει, έχουμε πιστήσει την προσοχή στο θέμα σε διάφορα πλαίσια. Για το κατά πόσο έχουμε κάνει αρκετά, αυτό είναι πάντοτε δύσκολο να το πω. Νομίζω πάντως πως η Ολλανδία ήταν μια από τις πιο δραστηριές χώρες όσον αφορά την προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα και στην Ολλανδική αντιπροσωπεία για τους κανονισμούς περί εγκρίσης τύπου έχουμε υποβάλει επανελειμμένως τα πορίσματά μας και πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα αυτά, τα πορίσματα αυτά ήταν και στη βάση της σχετικής νομοθεσίας. Οπότε ναι, ε, έχουν επιπτώσεις, έχουν επιπτώσεις όμως για τα αυτοκίνητα που θα κατασκευαστούν από εδώ και μπρο και όχι για αυτά που ήδη κυκλοφορούν. Μάλιστα, τελευταία μου παρατήρηση για την τελευταία σας διαφάνεια για την ποιότητα του αέρα στις πόλεις. Είπατε ότι λόγω των πολύ ψηλότερων εκπομπών των αυτοκινήτων στους δρόμους ποτέ δεν πρόκειται να πετύχουμε τα στάνταρ της ποιότητας του αέρα στις ευρωπαϊκές μας πόλεις. Το αναφέρατε αυτό και στην εκθεσή σας, στις εκθέσεις σας εδώ και χρόνια. Έχετε την αίσθηση ότι οι πολιτικοί ηθήνονται ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν κάνει αρκετά ή έχουν κάνει ελάχιστα για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα ενώ εστιάστηκαν περισσότερο στις τεχνικές προδιαγραφές για τα αυτοκίνητα και όχι στην ποιότητα του αέρα στις πόλεις. Uh, difficult question. <laughs> That's clear. Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την ποιότητα του αέρα γνωρίζουν όλα αυτά τα στοιχεία εδώ και καιρό. Δεν έχει σημασία το ότι πιστεύουμε εμείς. Σημασία έχει το ότι θεωρείται δεδομένο εδώ και αρκετό καιρό. Και ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει δοθεί αρκετή όθηση για να επιληθεί το θέμα. Αυτό δεν εξαρτάται όμως από εμά. Εμείς ε, το έχουμε γνωστοποιήσει, αλλά δεν έχει λάβει την απαραίτητη προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σμόκερς, άκουσα τα όσα είπατε. Έχω διαβάσει το υλικό που στείλατε. Έχω διαβάσει την, την έκθεσή σας και τη φετινή. Συνοψίζοντας, θα λέγατε με απλά λόγια ότι αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους για τις εκπομπές το Euro 6 τώρα. Έχουμε το διοξίδι του αζότου και το οξύδιο του αζότου. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητα. Το ντίζελ πέθανε ή μπορεί ένας κινητήρας πετρελαίου να κάνει τη δουλειά. Εγώ δεν, εμείς δεν νομίζουμε ότι πρέπει να καταργηθούν οι πετρελοκίνητοι τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητα για να επιτευχθούν οι στόχοι. Αυτό λέμε και στις απαντήσεις στις τεχνικές ερωτήσεις. Πιστεύουμε ότι με τις διαθέσιμες τεχνολογίες, εάν συνδυαστεί το EGR με το LNT, το ECR με κατάλληλο τρόπο και λειτουργήσει υπό διάφορες λειτουργικές συνθήκες, τότε τα πετρελοκίνητα οχήματα μπορούν να φτάσουν στη 8 ε, χιλιόγραμμα ε, ανά χιλιόμετρο. Είναι εφικτό δηλαδή αυτό. Σημαίνει πως αυτά τα οχήματα μπορούν να εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να ρηπαίνουν τόσο πολύ εφόσον φτάσουν σε αυτές τις επιδόσεις. Πολλά εκατομμύρια κόσμος ανέπνευσε αυτή τη στιγμή, αυτοί που κατασκευάζουν δηλαδή τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητα. Τώρα, εφόσον η τεχνολογία υπάρχει, τι πρέπει να αλλάξουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί και όλα σωστά η τεχνολογία αυτή. Αυτό που πρέπει να αλλάξει βασικά είναι ότι οι απαιτήσει, οι προδιαγραφές να είναι τέτοιε για την πλήρη λειτουργία του συστήματο. Γι' αυτό μιλάμε για το RDE. Το RD είναι καλή λύση με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλες οι προδιαγραφές. και θα καλύπτουν πραγματικές συνθήκες. Φυσιολογική οδήγηση δηλαδή και σε ποιο βαθμό όλα αυτά περιλαμβάνονται στη διαδικασία για το RD. Αλλά η αρχή της δοκιμής ε, στον δρόμο έχει πλέον αποδειχτεί Βλέπουμε ας πούμε ότι τα φορτηγά Euro 6 ε, για το οξύδιο του, α, του, του αζότου είναι καθαρότερα από ότι τα ε, ημιφορτηγά Euro 5, ακόμα και πιο καθαρά από επιβατικά αυτοκίνητα, γιατί ακριβώς οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες έχουν συμπεριληφθεί. Τρίτη μου ερώτηση. Αυτές οι τεχνολογίες ο συνδυασμό, δηλαδή αν χρησιμοποιηθεί καταλήλω, είναι ανταγωνιστικά, ανταγωνιστικές από άποψη κόστους σε σχέση με τις, ε, τους διζελοκινητήρες. Εξαρτάται από τι ορισμό θα δώσετε στο ανταγωνιστικό από άποψη κόστους. Το να προσθέσουμε τεχνολογία στο τα αυτοκίνητα να είναι πιο καθαρά, τα κάνει πιο ακριβά, αλλά δεν είναι αυτός ο χώρος να συζητήσουμε λεπτομέρειες του κόστους, αν πρέπει αυτό να επανεκτιμηθεί, εξπόστε θα χρειαστεί μια ειδική μελέτη. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ε, πρόβλημα της κότας και του αυγού όσον αφορά το κόστος αυτών των τεχνολογιών. Αν αυτές εφαρμοστούν σε πλήρη κλίμακα και παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα, θα μειωθεί και το κόστος. Εάν όχι, βεβαίως θα παραμείνει ψηλότερο Σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η ανταγωνιστική θέση των διζελοκίνητων σε σχέση με τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, αυτό επηρεάζει και το κόστος των ε, πετρελοκίνητων αυτοκινήτων. Το κόστος πάει, ε, αυξάνεται, αλλά αυτό είχε γίνει δεκτό ως τμήμα της νομοθεσίας Euro 6 με την ε, προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών. Υπάρχει χώρος για βελτίωση λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Dance. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ, δόκτωρα Σμόκερς, για την παρουσίαση που κάνατε. Εμένα με συναρπάζει αυτή η ιδέα του συνδυασμού τεχνολογιών και της ε, απόδοσης των αποτελεσμάτων που περιμένουμε. Είπατε ότι το, ένα κινητήρας CR δεν χρειάζεται κάποιο κουμπί για να σβήσει. Τώρα, για αυτές τις τεχνολογίες ιδιαίτερα όσον αφορά την λειτουργία του κινητήρα με τρόπο ώστε να μην βλάπτεται. Από ό,τι βλέπω κάποιοι κατασκευαστές, η Daimler ας πούμε, η οποία μειώνει την τεχνολογία κατά 5 βαθμούς, η Renault 17 βαθμούς. Ενώ η μέση θερμοκρασία στην Ευρώπη είναι 9 βαθμοί. Ποιος είναι ο μηχανολογικός λόγος γι' αυτό. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι και για μας οι κατασκευαστές μας δίνουν τις ίδιες εξηγήσει. Τεχνικώς είναι ε, λογική αυτή η εξήγηση. Η εφαρμογή της τεχνολογίας AGR, αυτό που λένε είναι ότι ότι το να σβήνει ο ψύχτης ε, ε, οδηγεί σε μικρότερη απόθεση καπνιάς μέσα στον κινητήρα. Αυτό από ό,τι φαίνεται οφείλεται στις, ε, ε, στη μικρότερη ε, εισχώρηση αέρα. Αλλά γύρω από το κινητήρα υπάρχει ένα σωρό θερμότητα. Ε, γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα του κινητήρα. Φαίνεται όμως να μην είναι τόσο τεράστιο αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό βασικά λέμε ότι με τα τωρινά συστήματα μπορεί να είναι πρόβλημα, αλλά σίγουρα δεν είναι αναπόφευκτο πρόβλημα ή άλλη το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεδομένων των όσων λέγατε νωρίτερα και των όσων περιλαμβάνονται στις γραπτές σας απαντήσεις, σε σχέση με τις, την ε, ενθερμό ε, το, το ξεκίνημα του κινητήρα Στη ΣΥΠΑ συμπεριλαμβάνουν την θερμό εκκίνηση στις διαδικασίες δοκιμών, ενώ στην Ευρώπη όχι. Δεδομένου ότι είπατε ότι η τεχνολογία EGR ειδικά θα έπρεπε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά σε υψηλές θερμοκρασίες. Για ποιο λόγο βλέπουμε ψηλότερες εκπομπές σε ψηλότερες θερμοκρασίες. Είτε δεν μας λέτε την αλήθεια που δεν το πιστεύω αυτό, είτε κάπου αυτή η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Υπάρχει άλλος λόγος για αυτή τη διαφορά. Εγώ νομίζω πως είναι το δεύτερο. Δεν είναι μόνο θέμα θερμοκρασίας. Αυτό που περιγράφω στο έγγραφο είναι ότι εάν κάνεις δοκιμές σύμφωνα με την νομοθεσία τύπου έγκρισης, ξεκινάμε με κρύα μηχανή, είναι ανάμεσα στις 20 και στις 30, στους 30 βαθμούς σημαίνει ότι μετά πρέπει να ζεσταθεί και ο υπόλοιπο κινητήρα και εκεί βλέπουμε ότι είναι ψηλέ οι εκπομπέ και μειώνονται όταν τα συστήματα θερμανθούν. Αν κάνουμε την ίδια δοκιμή, αλλά με μια, ένα κινητήρα που μόλι έχει σβήσει, είναι δηλαδή σε, στην κανονική θερμοκρασία λειτουργία τότε βλέπουμε ψηλότερε εκπομπές με θερμή και θερμό κινητήρα από ότι με ψυχρό κινητήρα. Αυτό αφορά το σημείο εκκίνηση, τι συνθήκη εκκίνηση του κινητήρα. Πρέπει να δούμε πού οφείλεται αυτό, αλλά αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουν οι κατασκευαστές. Πρέπει να είναι στη στρατηγική ελέγχου Πιστεύετε ότι οι δοκιμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θερμό, θερμή έναρξη του κινητήρα θα έπρεπε να γίνεται. Ναι, θα, θα μπορούσε. Δεν με eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφέρατε πολλά στοιχεία και βλέπουμε και από τις γραπτές απαντήσει ότι υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία τα οποία διευκρινίζονται περισσότερο. Τα πρότυπα οξυδίου του αζότου που είναι 18 mg ανά χιλιόμετρο μπορούν να επιτευχθούν με την τρέχουσα ε, τεχνολογία, οπότε δεν χρειαζόμαστε νέα τεχνολογία. Δεύτερον, αυτό δεν χρειάζεται να υπονομεύσει τη δουλειά που γίνεται για τι εκπομπέ διοξυδίου του άνθρακα. Μπορούμε να μειώσουμε και τα δύο. Τεχνικώ είναι δυνατόν. Στην πράξη, βέβαια, Ακόμα είμαστε μακριά από την επίτευξη αυτού του στόχου. Στην ερώτηση 2, πραγματικά ε, έχετε κάνει διάνα για το ζήτημα αυτό. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι ποιοι είναι οι λόγοι που συμβαίνει αυτό. Έχει να κάνει με το κόστος Μιλάτε για, την, το αυξημένο κόστος για κάποια ε, δυσδοκίνητα οχήματα και το χαμηλό περιθώριο κέρδους. Ε, θεωρείτε ότι αυτή μπορεί να είναι ε, ε, εύλογη εξήγηση. Πριν ακούσαμε ότι μιλούμε για 400 ευρώ αύξηση ανά ε, όχημα μετά από την κατάσταση των νέων συστημάτων δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το κόστος ε, των συστημάτων αυτών γιατί δεν το έχουμε μελετήσει λεπτομερώς. Αλλά αυτό που μπορώ να σας ε, πω και που είναι λογικό να το τεκμέρουμε είναι ότι το κόστος του συστήματο σε σχέση με το κόστος του οχήματο είναι πιο υψηλό. για τα μικρότερα οχήματα ε, παρά για τα μεγαλύτερα οχήματα, όπου εκεί τα περιθώριο κέρδου είναι πολύ μεγαλύτερο. Το ε, περιθώριο λοιπόν κέρδους ε, για το μικρό αυτοκίνητο ε, θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι για το μεγάλο. Αλλά επειδή δεν έχουμε κάνει ενδελεχή έλεγχο των, του κόστου των συστημάτων αυτών, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις τεχνικές τροποποιήσεις όμως. Ε, ουσιαστικά η RD πρέπει να κάνει το, την όλη δουλειά. Το θέμα είναι αν τα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε μπορούν να επιτευχθούν πιο γρήγορα με, ε, από ότι τώρα με τον τρόπο που γίνεται. Αν δηλαδή μπορεί να αλλάξει τώρα κάτι στα υπάρχοντα οχήματα, νομίζω ότι είναι δύσκολο να ε, εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο. Τα νέα οχήματα ίσως να μπορούν να επιτύχουν το στόχο αυτό, αλλά το ερώτημα μετά είναι πόσο γρήγορα μπορούν οι κατασκευαστές να αλλάξουν το σχεδιασμό των οχημάτων για να επιτύχουν γρήγορα το στόχο αυτό υπό συνθήκες πραγματική κίνηση. Ε, αυτό βεβαίω είναι ένα κομμάτι της συζήτησης. Και τι έχετε να μας πείτε για το, ε, για το επίπεδο φιλοδοξίας αυτών των δοκιμών RDA. Καταρχάς υπάρχει το θέμα του χρονισμού. Αυτό που ζητείτε είναι να είμαστε αποτελεσματικοί ε, σε πλήρες φάσμα. Και το άλλο είναι το θέμα της συμμόρφωσης. Και όπως είπα δεν είναι το θέμα μόνο συμμόρφωσης, αλλά και το σε ποιο βαθμό τον, την εφαρμόζουμε. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν περιθώριο αύξησης του επίπεδου φιλοδοξίας. Θα λέγαμε βεβαίως ότι μιλούμε για ε, συμβασμό. Θα μπορούσαμε να πάμε πιο γρήγορα, πιο έντονα, αλλά υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη για περισσότερα στοιχεία, για περισσότερε έρευνες που δεν έχουν γίνει ακόμα, οπότε χρειάζονται στοιχεία ε, για να δούμε τι μπορεί τελικά να επιτύχει η τεχνολογία, τι μπορεί να επιτύχει η βιομηχανία. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε ακόμα, γι' αυτό είναι δύσκολο. Στην απάντησή σας, στην ερώτηση 10, λέτε ότι τα PEMS ε, τα βλέπετε με επικριτική ματιά. Γιατί δεν, ε, μιλούμε, δεν ε, επικρίνουμε την εφαρμογή της τεχνολογίας PEMS. Είναι καλή αυτή. Αλλά υπάρχει και ένα επίπεδο ακρίβειας που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν καθορίζουμε ένα όριο με βάση, τα, ένα πρότυπο με βάση τις της PEMS. Υπάρχει μια βελτίωση σε σχέση με τα τρέχοντα συστήματα. Και υπάρχει και Το θέμα της ε, δυνατότητας να εφαρμόσουμε κάποιες από τις τεχνικές ε, ε, που μπορούν να επιτύχουν αυτήν την ακρίβεια. Η μέτρηση αυτή είναι τμήμα που ορίζει ακριβώς το κατά πόσο είναι ακριβές το σύστημα ή όχι. Θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των προδιαγραφών του συστήματος που ήδη ε, υπάρχουν. Η κυρία Μάισνερ, εκ μέρου του Άλτε. Ευχαριστώ. Δεν ήξερα ότι είμαι, ήταν η σειρά μου. Για τα PEMS. Μόλις ε, το συζητούμε, αναρωτιέμαι. Είπατε ότι Υπάρχουν δυνατότητε βελτίωσης φυσικά και κατά την άποψή σα, ποιε είναι αυτέ οι δυνατότητε βελτίωσης σε σχέση με το τι υπάρχει τώρα. Και άλλο ένα ερώτημα. Υπάρχουν εναλλακτικέ στα PEMS. Τα PEMS μέχρι τώρα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γιατί λέει κανεί ότι τα δεδομένα δεν είναι ακόμα ακριβή, αλλά εμά μα ενδιαφέρει πάρα πολύ ακριβώ αυτά τα δεδομένα να τα μετρήσουμε με την καλύτερη δυνατή τεχνολογία και όσο δυνατόν καλύτερα. Ποιε είναι λοιπόν οι δυνατότητε ε, βελτίωση που υπάρχουν και ποιε είναι οι εάν υπάρχουν. Uh, uh, Ευχαριστώ για την ανοχή σας. Δεν έχουμε προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος PEMS. Υπάρχει περιθώριο εξέλιξης, αλλά το θέμα είναι αν ε, χρειάζεται να το βελτιώσουμε και το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται τα όρια και πώς εφαρμόζονται οι μετρήσεις γιατί εδώ κυρίω μιλούμε για ε, παράγοντε συμμόρφωση. Το τρέχον πρόβλημα που έχουμε είναι ότι οι εκπομπέ σε πραγματικές συνθήκες ε, είναι 3, 4, 5, 6 φορέ υψηλότερε από τα συστήματα, από τα δοκιμέ έγκρισης τύπου. Ε, ήδη από, αν φτάσουμε το 1,5 σε σχέση με την έγκριση τύπου, έχουμε πολύ μεγαλύτερη βελτίωση. Οπότε τα PEMS μπορεί να είναι πολύ, λιγότερο, πολύ μικρότερο πρόβλημα όταν απαιτούμε 80 μιλιγκράμμα ανά χιλιόμετρο υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Οπότε η αξία των PEMS έχει να κάνει με, το, με την έκθεση τύπου που ήδη γίνεται και τις σχετικές δοκιμές. Βεβαίω εκεί υπάρχει ένα περιθώριο ερμηνεία. Και άλλη μια εξέλιξη που σα ανέφερα ε, είναι το σύστημα που έχουμε εμεί, το απλουστευμένο σύστημα μετρήσεων, και αυτό που θα μπορούσαμε να φανταστούμε είναι ότι κάνει κανείς μια αξιολόγηση σε διάφορες φάσεις, κάνει έναν έλεγχο από διάφορα είδη οχημάτων με βάση ένα μοντέλο για μια μεγάλη περίοδο σε συνθήκες οδήγησης, και βεβαίω εκεί υπάρχουν και οι συνθήκε, ε, οι καιρικέ, η θερμοκρασία. Οπότε το να μετρήσει κανεί μία μέρα μόνο δεν μα λέει πολλά. Και επίση βλέπουμε αν έχουμε αποτελέσματα εκτός των ορίων. Αν συμβαίνει αυτό, τότε μπορούμε να πάμε σε ε, μετρήσεις ευρέως φάσματος για να ερευνήσουμε τι ακριβώς μας λέει αυτό που έχουμε ε, μετρήσει, το αποτέλεσμα που έχουμε λάβει. Οπότε, τα PEMS μπορεί να μην είναι τόσο ακριβή για τις μετρήσεις στο εργαστήριο, αλλά το ερώτημα είναι αν θέλει κανείς να συντάξει μια, εκπονήσει μια ε, ε, νομοθεσία ε, που να μπορεί να ερμηνευτεί με τέτοιο τρόπο που να μην αποτελεί πρόβλημα το ότι δεν είναι ακριβή τα PEMS. Ωραία, δύο ερωτήματα επιπλέον. Μιλήσαμε πολύ για, το, για τη συμμόρφωση και βεβαίω ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο. Μιλάτε για 1,0 το οποίο θα είναι το καλύτερο. Από τα τεχνικά δεδομένα που έχουμε βλέπουμε ότι δεν είναι ε, δυνατό αυτό. Μα είπατε ότι όταν έχουμε 4, 5, 6 φορέ παραπάνω δεν είναι καλό, το 1,5 είναι καλύτερο. Μα είπατε εσεί, κατά την άποψή σα λοιπόν ποιο είναι πιο σκόπιμο, ποιο είναι πιο ρεαλιστικό. Δεύτερο ερώτημα. Μιλήσαμε για τα τζελοκίνητα και είπατε ότι δεν θα πρέπει να τα κατηγορούμε γενικώ, γιατί έχουν συμβάλει στη μείωση της, ε, των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα, αλλά το ερώτημα είναι, οι κινητήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν κίνηση θερμή ή ψυχρή, έχει σημασία το πώς ε, αλλάζουν οι εκπομπές τους. Δηλαδή έχει διαφορά, γιατί στην Ευρώπη έχουμε διαφορετικές ε, ε θερμοκρασίες και αυτό έχει προφανώς ε, επιπτώσεις και στις ε, εκπομπές. Για να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημά σας πρώτα, νομίζω ότι ακόμη και αν τα LNT, τα SCR εφαρμοστούν πλήρως σε αυτά τα σε αυτά τα οχήματα θα εξαρτάται πάντα η απόδοσή τους από, από τη θερμοκρασία και αυτό μάλλον θα έχουν να το αντιμετωπίσουν περισσότερο οι νότιες χώρες αλλά δεν θα είναι με, στο ίδιο εύρος που το βλέπουμε τώρα. τώρα, αν, αν φύγουμε από το, από το φάσμα των 20 με 30 βαθμών, ε, δεν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Στη Σκανδιναβία, ας πούμε, το χειμώνα τα, τα οχήματα θέλουν περισσότερο χρόνο για ε, θέρμανση παρά στις νότιες χώρες. Τώρα, για, τις, ε, για τη συμμόρφωση, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τη συμμόρφωση ένα δικό της περσέ κομμάτι γιατί έχουμε να κάνουμε με το πού εφαρμόζεται. Έχουμε να κάνουμε με την αξιολόγηση του, της δοκιμής, αν είναι στο, στο δρόμο το όχημα ή όχι. Περνάνε μέσα από ένα μοντέλο τα αποτελέσματα, καταλήγουμε σε ένα ε, αριθμητικό στοιχείο και πάνω σε αυτό βάζουμε τη συμμόρφωση και τους παράγοντες συμμόρφωσης. Και οπότε τα πράγματα ορίζονται από το φάσμα των συνθήκων οδήγηση που θεωρεί κανεί οι φυσιολογικέ αποδεκτέ. Ποιε είναι οι μετρήσει που, ε, αφήνει, που αφήνει λίγο στην άκρη κατά τη διάρκεια της, του υπολογισμού. Με βάση και το εργαλείο αξιολόγηση που έχουμε. Έχουμε λοιπόν μέσω αυτού του μοντέλου το αποτέλεσμα τον, το αριθμητικό στοιχείο πάνω στο οποίο εφαρμόζεται ο παράγοντα τη ε, ε συμμόρφωση. Ε, δεν είναι λοιπόν, ε, δεν έχει νόημα να χάσουμε τις, την, τα αποτελέσματα αυτά, γιατί η αξιολόγηση από, μέσα, από μόνη τη δεν μα λέει πολλά. Η κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούω την, ε, ε, τις εξηγήσεις σας. Στην, θα ήθελα να κάνω αρχίζοντας μία πολιτική ερώτηση. Η Fiat Chrysler λέει ότι τα οχήματά της πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Η εφημερίδα Bild αναφέρει όμως ότι αυτή η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικές διαφορετικές. Η, ε, η εταιρεία λέει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, ο Γερμανός Υπουργός παρενέβη και ότι θα πρέπει να αφαιθεί η εταιρεία στην ησυχία της, να κάνει τη δουλειά της. Έχετε κάνει κάποιε μετρήσεις για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και αυτό το software ε, που χρησιμοποιεί η εταιρεία αυτή, όντως ισχύει ότι το χρησιμοποιεί ή όχι. Uh, Ωραία, να ξεκινήσω το τελευταίο ερώτημα. Σε ποιο βαθμό τα οχήματα και οι κατασκευαστές που έχουμε ε, αξιολογήσει χρησιμοποιούν τέτοιες ε, συσκευές. Δεν ξέρουμε γιατί δεν το έχουμε ελέγξει. Δεν γνωρίζουμε. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι έχουμε κάνει δοκιμές ε, σε Fiat σειράς 5. Το είχαμε στο πρόγραμμα αξιολογήσεων το προηγούμενο έτος και όλα τα, ε, όλα δείγματα έδειξαν υψηλές ε, εκπομπές ε, στις, συνθήκε συνθήκες οδήγησης. Δεν μελετούμε όμως την χρήση τέτοιων συσκευών, οπότε δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι στην έκθεση αναφέρονται μόνο τα στοιχεία υπό συνθήκε οδήγηση. Τώρα για το πρώτο θέμα, για τη Fiat που λέει ότι τα οχήματα χρειάζονται την τρέχουσα νομοθεσία. Όλες, όλοι οι κατασκευαστέ το λένε αυτό. Και αυτό έχει να κάνει και με ένα ερώτημα που δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Δηλαδή, ποια είναι ακριβή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Λέει ότι τα οχήματα πρέπει να εφαρμόζουν μόνο τα πρότυπα που υπάρχουν για τι δοκιμέ ε, έγκριση τύπου. Πρέπει να υπονοείται κάτι τέτοιο ή λέγεται ρητά ή όχι. Πρέπει να τηρούνται τα όρια. Ε, είναι νομική νομίζω η συζήτηση αυτή περισσότερο και εμεί ω τεχνικοί εμπειρογνώμονε δύσκολα μπορούμε να την κατανοήσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι τη συζήτηση αυτό. Είναι καλό το ερώτημα, αλλά δεν έχω απάντηση. Ούτω ή άλλως θα επανέλθει το ερώτημα αυτό και σε άλλες ε, συζητήσει. Ναι, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ε, συμφωνώ. Συμφωνώ με αυτά που είπατε και με όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, όπου προσπαθήσαμε να καταρτήσουμε κάποιους ε, κανόνες και πλέον έχουμε φτάσει ε, σε μια κατάσταση όπου πραγματικά έχουμε ρεζιλευτεί. Ε, ορίσαμε δηλαδή οριακές τιμές οι οποίες προφανώς και δεν τηρούνταν από την αυτοκινητοβιομηχανία. Και είπατε εδώ ότι τα PEMS δεν σχετίζονται ακριβώς με αυτό το θέμα διότι ε, δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβούς μέτρησης των δεδομένων και ότι θα πρέπει η νομοθεσία να προβλέπει και άλλες προϋποθέσεις εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι μπορούμε να καθορίσουμε κανόνες οι οποίοι να είναι και υλοποιήσιμοι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι απαντήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα συμμεριζόμαστε τις παρατηρήσεις παρατηρήσεις ότι έως σήμερα η νομοθεσία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ότι οι εκπομπές θα είναι όσο το δυνατόν ε, χαμηλότερος. Αν κατάλαβα καλά τη διερμηνία, είπατε ότι ε, η μέθοδος PEMS δεν θα είναι, ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα. Εμείς δεν είπαμε αυτό. Αντιθέτως, το PEMS, η μέθοδος PEMS είναι μια πολύ χρήσιμη ε, ε, μεθοδολογία, αλλά από την άλλη ε, είναι αλήθεια ότι ε, βρίσκονται, ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των πραγματικών και των εργασιακών συνθήκων. Αλλά αν αξιοποιηθεί σωστά ο εξοπλισμός αυτός, τότε μια χαρά ε, μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Είπατε ότι η νομοθεσία ε, είναι κάπως ασαφής όσον αφορά τις, τις συσκευές αναστολής. Αν δείτε όμως τι λέει η νομοθεσία, αναφέρεται ε, ότι τα πρότυπα θα πρέπει να τηρούνται υπό κανονικές συνθήκες. Απαγορεύονται οι συσκευές αναστολής, οι διατάξεις αναστολής, εκτός αν μια τέτοια διάταξη είναι απαραίτητη για να προστατευτεί ο κινητήρας από ατυχήματα ή ε, βλάβη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του οχήματος. Αυτό είπατε ότι μπορεί να εξασφαλιστει η ασφαλης λειτουργια του οχηματος αυτο ειπατε οτι μπορει να συσχέει για συγκεκριμένο αριθμό και για συγκεκριμένο τύπο ε, ε, οχημάτων. Εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε αυτές οι συσκευές αναστολής να απαγορεύονται για όλα τα είδη οχημάτων. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε νομικές αρμηνίες για το κείμενο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, όποτε το έχουμε συζητήσει με διάφορους ε, ενδιαφερόμενους, ακούμε διάφορες ερμηνείες, διάφορες απόψεις. Εμείς δεν είμαστε νομικοί. Ε, τώρα είναι δύσκολο για μας το, το θέμα. Γι' αυτό και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το να πούμε ότι χρησιμοποιήθηκαν συσκευές αναστολής. Ωραία, εντάξει, άρα δεν θα σας πειράξω. Αν και, θα, θα, μπορούσατε να, θα μπορούσατε να πείτε ότι ε, είναι ασαφής ε, η διατύπωση της ομοθεσίας για εσάς, όχι ότι είναι γενικά ασαφής. Μπάς περιπτώσει, όταν το 2010 είχατε κάποια απορίσματα, κάποια αποτελέσματα, αλλά και το JRC είχε εντοπίσει πολύ υψηλές εκπομπές, τι συνέβη τότε μεταξύ του TNO και του JRC. Φαντάζομαι ότι θα διοργανώσατε κάποιες ε, συναντήσεις, δεν μπορεί. Yes, uh, thank you for this question. Um, Ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό. Φυσικά κάναμε πάρα πολλές συναντήσεις με το Κοινό Κέντρο Έρευνας, αλλά όχι σε διμερή βάση. Τόσο το JRC όσο και το TNO συμμετείχαν στο πλαίσιο διαφόρων ομάδων εργασίας ε, και ε, κοινοποίησαν τα ευρήματά τους για τις πολύ ψηλές εκπομπές. Αυτές οι πληροφορίες λοιπόν δημοσιεύτηκαν και τέθηκαν στη διάθεση όλων των ενδιαφορομένων μερών. Ε, εξ όσων γνωρίζω, Αυτά γνωρίζον, ήταν γνωστά ήδη από το 2010 και κάποια εθνικά Ινστιτούσα είχαν, Ινστιτούτα είχαν απαντήσει τότε ότι οι μετρήσει αυτές δεν είναι σωστές. Ισχύει. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Συγγνώμη, δεν το θυμάμαι αυτό. Τι να κάνουμε. Πάντω, είναι αλήθεια ότι το 2010 και 2011 έγιναν συναντήσεις επί, επί αυτών των θεμάτων. Οπότε αν εσείς δεν θυμάστε, μπορείτε τουλάχιστον να μας πείτε γιατί δεν έγιναν και τόσα πολλά πράγματα μετά τις ε, συνεδριάσεις αυτές. Δηλαδή μιλώ για νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν ανελήφθησαν ποτέ, η Κομισιόν ήταν εκεί. Με βάση τα δικά σας πορίσματα και ευρήματα θα περίμενε κανείς ότι θα είχαν αναλυφθεί δράσεις άμεσα. Ε, συγγνώμη, ε, δεν ε, εναπόκειται στο τι TNO να κρίνει γιατί δεν έγινε αυτό. Εμείς, εμάς ο ρόλος μας είναι συγκεκριμένος σε αυτές τις ομάδες και αυτό που κάνουμε είναι να κομίζουμε ανεξάρτητες πληροφορίες όσον αφορά τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες. Τώρα το τι κάνουν οι άλλοι δεν είναι δικό μας θέμα, ούτε θα αναλάβουμε εμείς την ευθύνη. Ναι, τα, τα, ακόμα και στα νομικά ζητήματα, τα, τα πολιτικά ερωτήματα... Ε, ναι, ναι, ξέρω, αλλά οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν σε αυτές τις ε, συνεδριάσεις και γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα και η δική τους παρουσία. Ωραία, να ξαναπεράσουμε στην, ε, στη θερμή και στην ψυχρή εκκίνηση. Ξέρουμε ότι στις ΙΠΑ τα αποτελέσματα είναι ακριβώς αντίθετα, ανάποδα. Ε, που είναι και λογικά ε, αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική, αυτά που μετρώνται στην Αμερική. Στην Ευρώπη πάλι έχουμε ε, ε, τις, τα, τις αντίθετες μετρήσεις και τα αντίθετα αποτελέσματα. Απάντηση. Ε, αυτό είναι νέο για μένα. Πρέπει να, το, να, να δούμε περί τίνος οχήματος πρόκειται, πιο ε, όχημα κάθε φορά, αν χρησιμοποιήθηκαν συσκευές αναστολής, διατάξεις αναστολής. Ε, είναι πάντως, όπως είπατε, λογικό οι εκπομπές να είναι υψηλότερες σε ψυχρή εκκίνηση παρά σε θερμή εκκίνηση. Αν ε, υπάρχουν τέτοια ευρήματα, τότε φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπήρξε χρησιμοποίηση συσκευών διατάξεων αναστολής. Α, κάτι τέτοιο πάντως ε, είναι πολύ δύσκολο να το κρίνει κανείς. Ε, μπορείτε να μας δώσετε την απάντησή σας γραπτός, λέει η Πρόεδρος. Με το, να, να έχετε και τον χρόνο που χρειάζεστε για να δώσετε μια ολοκληρωμένη απάντηση. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις που έχετε δώσει μέχρι τώρα. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του παράγοντα συμμόρφωσης. Με βάση τις απαντήσεις σας στην ερώτηση 1, είναι προφανές ότι δεν πρέπει να αναμένουμε νέες εξελίξεις και νέες ε, τεχνολογίες για να μειώσουμε το οξύδιο του αζότου εφόσον αυτές που υπάρχουν λειτουργούν όταν χρησιμοποιηθούν σωστά και συνδυαστούν σωστά. Πιστεύετε ότι ένας παράγοντας συμμόρφωσης ε, που εφαρμόζεται στα όρια του νόμου, όπως ορίστηκα το 2,1 μέχρι το 2020, μπορεί να είναι αιτιολογημένο. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα σωστά, με ρωτάτε πώς κρίνουμε την καταλληλότητα των ε, συντελεστών συμμόρφωσης όπως αυτοί έχουν επιλογή, επιλεγεί. Όπως είπα και πριν, η αυστηρότητα αυτών των ε, συντελεστών εξαρτάται από τον αριθμό στον οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής και αυτό εξαρτάται με τη σειρά του από το ποιες μετρήσεις θεωρούνται έγκυρες και όλα αυτά ακόμα βεβαίως βρίσκονται υπό συζήτηση. Οπότε δεν μπορούμε να τα εξετάσουμε ξεχωριστά αυτά τα ζητήματα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και παρότι παρουσιάστηκαν στον τύπο οι, οι συντελεστές συμμόρφωσης αυτή ως μια επιτυχία της αυτοκινητομηχανίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς ελπίζουμε ότι θα ε, καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα τελικά. Αλλά όπως είπα οι συντελεστές αυτοί είναι μία μόνο μεταβλητή της ε, εξίσωσης. Δεν θα πρέπει να επικεντρώνουμε μόνο στους συντελεστές, θα πρέπει να εξετάζουμε ολόκληρη τη διαδικασία σε συνεργασία με τον κατασκευαστή και ε, η νομοθεσία θα πρέπει να είναι επαρκώς αυστηρή ώστε τα επόμενα χρόνια να παρακολουθούμε τα οχήματα και τις ε, εκπομπές τους σε πραγματικές συνθήκες. Γιατί εξ όσων γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή η νομοθεσία δεν προβλέπει τίποτα για τις ε, μετρήσεις πραγματικών συνθήκων. Γιατί αν γίνουν οι μετρήσεις τόσο σε εργασιακό επίπεδο όσο και σε πραγματικές συνθήκες, τότε μπορεί κανείς να συγκρίνει. Κατανοώ αυτό που λέτε. Αλλά πώς πιστεύετε ότι αυτό θα εξασφαλίσει την ε, τεχνολογική ουδετερότητα. Λαμβάνοντας και υπόψη ότι οι συντελεστές συμμόρφωσης αυτοί έχουν, ε, έχουν θεσπιστεί μόνο για τα τζελοκίνητα οχήματα. Δεν νομίζω ότι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή η τεχνολογική ουδετερότητα. Αντιθέτως, το RDE στην ουσία διορθώνει την ομοθεσία και την επαναφέρει στον αρχικό της στόχο. Ε, κατά την ε, εκπόνηση του Euro 6 θεωρήθηκε ως δεδομένο ότι ε, οι τεχνικές μέθοδοι μέτρησης θα εξασφάλιζαν ότι οι μετρήσεις ανταποκρίνονται στις συνθήκες πραγματικής οδήγησης. Διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι και είδαμε ότι το RDE τελικά είναι διαφορετικό από το, από αυτό που συμβαίνει στον ε, πραγματικό κόσμο. Στην πραγματικότητα λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια διόρθωση της νομοθεσίας. Και αν το Euro 6 είχε γίνει αποδεκτό ως ε, μια, ένα λογικό μέτρο ε, από την Κομισιόν, από το Κοινοβούλιο, τότε ε, δεν έχετε εσείς κάποιο πρόβλημα, δεν θα έπρεπε να έχετε κάποιο πρόβλημα, διότι το RDE δεν κομίζει κάτι νέο, ούτε, ούτε προσθέτει κάποιο στοιχείο, ίσα ίσα εξασφαλίζει τον, ότι θα επιτυγχάνετε ο στόχος που είχατε εσείς θέσει με το Euro 6. Κύριος Τσόγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ παρόντε. Όπω ε, λέτε στην εισαγωγή στι απαντήσει οι εκθέσει ε, που ε, δημοσιεύθηκαν φέτο από το ΤΙΟΝΟ δείχνουν απόκληση ανάμεσα στι εργαστηριακέ εκπομπέ μονοξιδίου και τι εκπομπέ υποπραγματικέ συνθήκε. Ε, Τρει με πέντε φορέ πιο υψηλέ ήταν οι εκπομπέ και αυτό ο παράγοντα μου πολλαπλασιάζεται από 10 σε 20 σε περίπτωση επιτάχυσης ή γρήγορη. Οδήγησε Αυτό είπατε ότι οδήγησε σε ιδιαίτερε αντιδράσει όσον αφορά ε, μια αναπάτη ή κάποια συσκευή αναστολής. Πώς εξηγείται μια τόσο σημαντική απόκληση πριν από τις ε, αποκαλύψεις του περασμένου Σεπτεμβρίου ή η κοινή γνώμη θεωρούσε ότι αυτή η απόκληση ήταν ε, μοιραία και ότι οφιλότερο στην συμπεριφορά του οδηγού ε, βλέπουμε ότι οι δικές σας απαντήσεις έχουν άλλο περιεχόμενο. Εσείς λέτε πως οι κανόνες 06 ε, αφορούν τον περιορισμό των εκπομπών μονοξιδίου, ε, οξυδίου του αζότου, αλλά και ότι γίνεται να συνδυαστεί η μείωση εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα και οξυδίου του αζότου φαίνεται να περάσατε από μια κάποια ανοχή σε έναν ανεφόρον, μια ανεφόρον αισιοδοξία. Ε, ε, δεύτερη ερώτηση, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτή την εξέλιξη. Και τέλος φέρετε να, επίσης να λέτε ότι όλες οι τεχνολογίες μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά ώστε να περιοριστούν οι ρήποι και ότι ο, η τεχνολογική πρόοδος είναι μόνο ένας ε, ενάρετος κύκλος. Όμως, όταν μιλάμε για περιορισμό του σχηματισμού του οξυδίου του αζώτου, περιορίζονται η αποδοτικότητα του κινητήρα μειώνοντας την καύση. Πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης του καυσίμου. Έχετε εκτιμήσεις για το κόστος αυτών των ε, καινοτομιών για τον καταναλωτή και κατά πόσο είναι βιώσιμα αυτά τα νέα αξεσουάρ όσον αφορά την κατασκευή τους και τη συντήρησή τους. Ευχαριστώ που θα μου απαντήσετε σε κάθε μια από αυτές τις ερωτήσεις. Ελπίζω να θυμάμαι τα, τις ερωτήσεις σας. Να ξεκινήσω αυτή τη φορά με την πρώτη ερώτησή σας. Νομίζω ότι αυτό που είπατε είναι ότι είναι φυσικό να περιμένει κανείς ότι οι εκπομπές θα είναι υψηλότερες όταν ο κινητήρας καταπονείται περισσότερο, όταν επιταχύνει για παράδειγμα. Ε, Φυσικά, υπό ορισμένε συνθήκε οι εκπομπέ είναι υψηλότερε, υπό πιο αντίξιο ε, συνθήκε οι εκπομπέ είναι υψηλότερε από ότι όταν οι συνθήκε είναι πιο ομαλέ. Το ζήτημα που μας απασχολεί είναι αν είναι διαφορετική, ε, αν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ε, εργαστηριακών και των πραγματικών εκπομπών. Ε, βλέπουμε ότι οι πραγματικές εκπομπές είναι πολύ ε, υψηλότερες και κάτι που το επιβεβαιώνει αυτό είναι ότι όταν εξετάζουμε, όταν ε, ελέγχουμε οχήματα σε πραγματικές συνθήκες, σε αντίξωες όμως πραγματικές συνθήκες, πάλι οι εκπομπές είναι υψηλότερες από ότι όταν το φορτίο κινητήρα στην δοκιμή στην εργαστηριακή είναι υψηλή. Είναι, είναι υψηλό. Αυτό... Το να υπήρχε μια ποσοστιαία μεταβολή ε, μεταξύ των μετρήσεων, αυτό θα ήταν αποδεκτό. Αλλά το να είναι διπλάσιες, τριπλάσιες έως και εξαπλάσιες οι μετρήσεις, ε, αυτό δεν μπορεί να, να συμβαίνει συμπτωματικά ούτε οφείλεται απλά στην ε, διαφορά των ε, πραγματικών συνθήκων. Ε, αν δείτε λοιπόν ότι αν δείτε λοιπόν έναν κινητήρα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι πάντοτε ευθύγραμμη η αύξηση των εκπομπών με την αποδοτικότητα, με, την, με το φορτίο του κινητήρα αν το, το ότι υπάρχει ένα after treatment δηλαδή των εκπομπών στην ουσία μπορεί κανείς να ε, επιτύχει μείωση ε, των διοξιδίων, του, του διοξιδίου του άνθρακα και άλλων ε, ρηπογόνων αερίων. Φυσικά όλα αυτά είναι δαπανηρά και θα χρειαστεί να εγκατασταθεί ε, σχετική τεχνολογία. Ε, η πρόεδρος λέει ευχαριστώ πολύ, όλοι πήρατε ένα λεπτάκι από τη σημαία. Ε, δεν θα μπορέσω να σας το δώσω αυτό στο δεύτερο κύκλο συζητήσεων, ερωτήσεων, δεν θα τα καταφέρουμε. Είναι ένας συντελεστής συμμόρφωσης και αυτός. Θέλω τα ερωτήματα να είναι σαφή και οι απαντήσεις όμως να είναι σαφείς και δεν θα επιδείξω τόση ανεκτικότητα όσο ε, έδειξα στην, ε, πρώτη, στον πρώτο γύρο συζητήσεων. Ο eigenlijk aan onze verwachtingen en is wat we verhoopt hebben. En zet uh, uiteraard de constructeurs ertoe aan om hè, belangrijk... Is Ο συμβιβασμό στον οποίο κατέληξε το Κοινοβούλιο στην ουσία ανταποκρίνεται και σε αυτά που εμείς περιμέναμε να δούμε. Ε, δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη η στόχη. Especially if the the details are implemented in right way, will uh, make sure that manufacturers... Με το σωστό τρόπο θα πρέπει οι κατασκευαστές να μεριμνήσουν ώστε οι εκπομπές ε, στους δρόμους να είναι πιο ε, συμμορφούμενες προς τα όρια. Ο βαθμός στον οποίο ε, θα εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις RDE και δημιουργούν δυναμική όπου οι πρώτοι θα ανταμυφθούν, ε, αυτό είναι αμφίβολο, γιατί υπάρχει ένα αδιέξοδο, γιατί θα πρέπει οι πρώτοι να αποδείξουν στους υπόλοιπου ε, υπόλοιπους κατασκευαστές ότι ήταν καλύτεροι. Μήπως έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα το, το δίλημα του, του, του, αυτό του φυλακισμένου. Μήπως οι πρώτοι όντω θα πρέπει να αναμειχθούν γιατί αυτό βοηθά οτιδήποτε υπάρχει διαθέσιμο να λυθεί δείχνει μάλλον ότι οτιδήποτε είναι ήδη διαθέσιμο, ε, βοηθά στο να λυθούν τα προβλήματα των πόλεων. Ναι. Αναφερθήκατε στο e σε πρόγραμμα ελέγχου των εκπομπών και το ΣΕΜΣ, το ΣΕΜΣ, το σύστημα αυτό, είναι ένα πρόγραμμα δεύτερης γενεάς. Όχι, να σας πω, δεν είπα ότι το ΣΕΜΣ είναι ανακριβές, γιατί αυτό φάνηκε να προτείνεται. Η ακρίβεια του ΠΕΜΣ, εξορισμού είναι μικρότερη από ό,τι τα μεγάλα συστήματα που μπορεί να έχετε σε ένα εργαστήριο, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο πρόβλημα, γιατί υπάρχει χώρος πάντα για βελτίωση. Όσον αφορά το σύστημα ΣΕΜ δεν νομίζω πω εδώ πρέπει να κάνουμε διαφήμιση για το δικό μα σύστημα. Πρόκειται για ένα απλοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί και κάποια σήματα από το αυτοκίνητο. Και γι' αυτό τον λόγο έχει χαμηλότερη ακρίβεια από ό,τι το πέμψε θεωρητικά, ενώ στην πράξη βλέπουμε πολύ καλή αντιστοιχεία ε, των μετρήσεων στο εργαστήριο και των μετρήσεων με το πέμψε. αλλά τουλάχιστον είναι πολύ καλή συσκευή ελέγχου, screening, ε, ανάλογα με τα άλλα αποτελέσματα, μέτρηση πούμε, αυτοκινήτων για μια ολόκληρη χρονιά στους δρόμους, να δούμε αν είναι όντως αυτοκίνητα που λειτουργούν με τον τρόπο που πρέπει. Αλλά όπως σας είπα, εδώ δεν πρέπει να κάνω διαφήμιση εγώ για την ανάπτυξη. Κυρία Μποναφέ. Δεν είναι η κυρία Μποναφέ, δεν ακούσαμε το όνομα. Ε, λέτε ότι τα συστήματα παραπληρωματικά ε, για τη μείωση διοξιδίου του άνθρακα και οξυδίου του αζότου μπορούν να λειτουργήσουν χωρί να δημιουργήσουν πρόβλημα στου κινητήρε. Σε πολλέ προηγούμενε ακούσαμε ότι η παρουσία τη σύνδεση δυο δύο-τριών τεχνολογιών κατά τη ε, ρήπανση για το ε, οξύδιο του, ανθρώπου, του αζότου θα επέτρεπαν να μείνουμε κάτω από τα όρια. Μήπω λοιπόν θα είναι καλό να μπουν και στα ευελαφριά οχήματα δύο συστήματα για το οξύδιο του αζότου ενώ θα τηρείται η τη λειτουργία του κινητήρα. Καταρχά. οι τεχνολογίε θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ουδέτερε. Να ορίσουμε δηλαδή στην ε, νομοθεσία τι θέλουμε ω επίδοση και όχι τι θέλουμε ω τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί. Γιατί η συνοχή, η συνέπεια, η διαλειτουργικότητα ε, πρέπει να δούμε ε, αν καταρχήν ε, υπάρχει λόγο το, με βάση το αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί αλλά και με βάση το λογισμικό με βάση το οποίο λειτουργούν αυτές τις τεχνολογίες. Να δούμε δηλαδή αν αυτά τα συστήματα λειτουργούν με τρόπο ώστε να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και έπειτα να δούμε και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου, τι εκπομπέ έχει και μετά να δούμε τι βάζουμε πάνω μόνο σαν τεχνολογία. Μια άλλη ερώτηση, πάντα στην πλαίσιο της πρώτης ερώτησης. Μιλάτε για απόθεση καπνιάς που μπορεί να βουλώσει το σύστημα. Αλλά είπατε ότι δεν μπορέσατε αυτό να το επαληθεύσετε, να το εξακριβώσετε. Δηλαδή προσπαθήσατε να ξανακάνετε αυτό το πείραμα, αλλά πετύχατε. Και εν γέννη τι σημαίνει κατά τη γνώμη σας το, επιχείρημα της προστασίας του κινητήρα και πώς ε, οι συσκευές κατά της ρήπανσης μπορεί να βλάψουν ε, τον κινητήρα. Συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι μια ερμηνεία μιας απάντησης που έδωσα ήδη. Η σημερινή ερμηνεία είναι ότι όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές μπορεί να ε, χαλάσει ο κινητήρας. Μπορούμε όμως αυτό να το διορθώσουμε ε, θερμαίνοντας τον αέρα με τη, με τη θερμότητα του κινητήρα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε γιατί δεν έχουμε αναπτύξει κάποιο σύστημα, δηλαδή δεν το έχουμε δοκιμάσει στην πράξη. Αλλά θα μπορούσαμε όντως να κατευθύνουμε τον αέρα μέσα από τον κινητήρα ώστε να θερμανθεί επαρκώς. Πιστεύουμε πάντως πως είναι εφικτό αυτό από τεχνικής άποψης. Η κυρία Γκροστέτ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη σας, είναι τα, τα νέα όρια εκπομπών, ΕΡΟ 5 και ΕΡΟ 6, έχουν ε, ε, περάσει αρκετά μακρές ε, μεταβατικές περιόδους ώστε να εφαρμοστούν σωστά. Και έπειτα, τι γίνεται στην Ιαπωνία ή στις ΗΠΑ. Ε, last question first again, uh, but without an answer because I don't really, uh, I'm not in a position to comment on. Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω την ε, Αμερικανική ή Ιαπωνική νομοθεσία γιατί δεν τη γνωρίζω επαρκώς. Τώρα, αν ε, το ΕΡΟ 5 και το ΕΡΟ 6 πέρασαν αρκετά μακρά χρονική μεταβατική περίοδο, από ό,τι γνωρίζω οι προδιαγραφές είχαν διοριστεί το 2005, αν δεν κάνω λάθος και άρχισαν να εφαρμόζονται το 2005 ή Πρέπει να το ψάξω μισό λεπτό. 2009. Ε, 2009, δηλαδή τέσσερα χρόνια ε, μεταβατική περίοδο για το Euro 5 και 8-9 για το Euro 6. Πιστεύουμε ότι είναι επαρκής χρόνος ως μεταβατική περίοδος. Άλλη ερώτηση. Το Κοινοβούλιο μα εργάζεται επί προτάσεως τη ε, βιομηχανία για να βελτιωθεί το σύστημα έγκριση διοδότηση των οχημάτων. Κατά τη γνώμη σα, αυτό μπορεί να επιτρέψει στην κάλυψη των ε, ισχυών των ε, κενών νομικών κενών. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από τις απαιτήσεις που προστίθεται στις δοκιμές ε, έγκρισης τύπου αλλά βεβαίω θα πρέπει να προσέξουμε όλε τι λεπτομέρειε γιατί τελικά η αποτελεσματικότητα και η αυστηρότητα εξαρτώνται από την πρακτική. Όλε τι διαδικασίε για τι διάφορου δοκιμέ και τα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα σημείο που δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε καμιά ανησυχία. Είναι κάτι που θα χρειαστεί να προσέξουμε. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μένα τώρα και δεν χρειάζεται να μπω εγώ τώρα σε λεπτομέρειε πολιτικέ για ένα θέμα που είναι υποσυζήτηση. Ο κ. Να επανέλθουμε στο θέμα της θερμοκρασίας. Γιατί υπήρξε ένα είδος... Ε, ε, υπήρχε μια ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε εσά και τον κύριο Εκχάουτ πριν από λίγο. Θέλω απλά να καταλάβω καλά. Η αιτιολόγηση μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει κάτι που σβήνει τις τεχνολογίες αναστολής. Αυτό λέτε, ο κρύος αέρας Απλά θέλω να μου το καταλάβω. Λοιπόν, και πάλι δεν κατάλαβα τι εννοείται ψηλέ θερμοκρασίε. Δοκιμή ψυχρή, ψυχρό κινητήρα, σύμφωνα με τη διαδικασία. Όλος ο κινητήρας δηλαδή να είναι στους 20 με 30 βαθμούς, αυτό που, μιλά, αυτό που καλούμε κρύο κινητήρα, ενώ ο θερμός κινητήρας είναι στους 80 με 90 βαθμούς. Ένας κινητήρας που ήδη έχει λειτουργήσει για κάποια ώρα. Έχουμε το παράδειγμα των διαφόρων κατασκευαστών που έβαλαν σε λειτουργία ε, το, τις συσκευές μετά τους 30 βαθμούς δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο ε, κύριος Δάνος, απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις, είπατε ότι η θερμοθερμοκρασία, η εξωτερική και το προσχετικό πράγμα μπορούν να ξεπεραστούν θερμάνοντας τους κινητήρες. Στη ΣΥΠΑ έχουν μείον 4 βαθμούς όσον αφορά την προστασία του κινητήρα. Στην Ευρώπη έχουμε 5, 10... Μέχρι και 17 βαθμούς ε, χαμηλότερα. Γιατί Εάν μείον μία-τέσσερα βαθμοί είναι η σωστή δοκιμή, μπορείτε ότι και αυτό μπορεί να ανασταλεί μέσω της θέρμανσης του αέρα που εισέρχεται στο κινητήρα. Ναι, να σας πω ότι η νομοθεσία, είπα, είναι στοχευμένη προς άλλα οχήματα, γιατί το, ε, ε, οι διζελοκινητήρες είναι ένα μυστήριο φαινόμενο στη ΣΥΠΑ και όλα τα όρια ε, αναφέρονται σε όρια που μπορούν να πετύχουν οι διζελοκινητήρες. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει εδώ να συζητήσουμε αν, είναι μείον 4, 0 ή 4 συμβαθμοί. βαθμοί. Αυτό που έχει σημασία είναι αν η νομοθεσία ζητά από τους κινητήρες να συμμορφώνται προς τις, κανονικές, τις εκπομπές κανονικών συνθηκών. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Όταν μιλάμε για κανονικές συνθήκες θα πρέπει να είναι ε, συνθήκες που ισχύουν συχνά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δοκιμές να γίνονται κάτω από κανονικές συνθήκες και μείον 10 βαθμοί Κελσίου είναι φυσιολογική φυσιολογικές συνθήκες. Μείον 5, μείον 10 είναι λογική η θερμοκρασία και αν είναι αυτό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, αυτό είναι λεπτομέρεια. Χένκελ. Yeah, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην παρουσίαση σας είπατε ότι μεταξύ του γύρω 1 και του γύρω 5 και, του εκπο, και τους ε, εκπομπές αυτών των ε, οχημάτων η, τα αριθμητικά στοιχεία είναι σταθερά. Ε, και είδαμε και αρκετά επιθετικούς στόχους. Αν καταλαβαίνω σωστά τα στατιστικά στοιχεία, η διαφορά μεταξύ του, των πραγματικών συνθήκων και του στόχου αυξάνεται. Ερώτημα λοιπόν από την επιχειρηματική κοινότητα. Αν ε, υπάρχουν πολύ επιθετικοί στόχοι, συνήθω ε, κανείς δεν προσπαθεί και το αποτέλεσμα είναι τελικά το αντίθετο. Δεν θα ήταν λοιπόν καλύτερα να επικεντρωθούμε στην επίτευξη ας πούμε του Euro 5 αντί να καταλήξουμε στο Euro 6 και να πούμε ότι τελικά διευρύνεται το χάσμα. Και τι γίνεται αν πούμε τώρα ότι θέλουμε να έχουμε και το Euro 7 και το Euro 8. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι απλό. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να επικεντρωνόμαστε στην, επί... στην επίτευξη κάποιων στόχων ή είναι πιο σημαντικό να θέτουμε όλο και καινούριου στόχους. Και οι δύο στόχοι τέθησαν ε, την ίδια χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίω ε, και τα χρονικά όρια και τις δυνατότητες που υπήρχαν. Όταν λοιπόν ε, τέθησαν τα πρότυπα γυρω 5, 6, με βάση τις αξιολογίες που είχαμε κάνει τότε, είχαν θεωρηθεί εφικτά με την διαθέσιμη τεχνολογία που είχαμε, με την προπόθεση ότι θα εφαρμοστεί η τεχνολογία αυτή με την απαραίτητη τεχνογνωσία και με τον σωστό τρόπο. Ε, θεωρούμε ότι όντω εφαρμόζεται η τεχνολογία, αλλιώ ε, δεν θα είχαν επιτύχει τα αποτελέσματα αυτά, τα οχήματα, όταν πέρασαν από τι διάφορε δοκιμέ, θα είχαν αποκλίνει από, την, ε, από τα πρότυπα. Και όπως Έδωσα και προηγουμένω απαντήσει σε πιο τεχνικέ ερωτήσει. Θεωρούμε ότι η τρέχουσα τεχνολογία είχε σκοπό να εφαρμοστεί το γύρο 5 και το γύρο 6 και να οδηγήσει σε αποδεκτά όρια εκπομπών σε ένα πιο ευρύ φάσμα, ε, σε ένα πιο ευρύ φάσμα ε, λειτουργουσών συνθήκων. Ε, θεωρούμε ότι με την τεχνολογία που έχουμε έχει καταστεί δυνατό να επιτύχουμε τους στόχους, αλλά τελικά με την νομοθεσία που υπάρχει τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που είχαμε επιθυμήσει από την αρχή. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα η σωστή στιγμή να, να συζητήσουμε την ε, σκοπιμότητα των στόχων. Και αν γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εξπόστα αξιολόγηση εκ των υστέρων για να συλλέξει κανεί καλέ ε, πληροφορίε και να έχει μια σωστή συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν τώρα να το συζητήσουμε αυτό. Ναι, αλλά φαίνεται ότι είναι αρκετά ευρεία η πρακτική αυτή της προσπάθειας επίτευξης στόχων με μεθόδους που δεν είναι αποτελεσματικές. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα εγώ έμαθα ότι δύο ιαπωνικές κατασκευάστες εταιρείε. Ε, ασχολούνται κυρίως με το hardware και όχι το software. Ε, δύο, δύο άτομα παρετήθηκαν από, την, από τις θέσεις τους διότι ο ένας παρουσίασε ε, οχήματα που ήταν πιο ελαφρά από, την, από, τα, από το ότι επιτρεπόταν. Έχετε κάποια αντίστοιχη εμπειρία. Συγγνώμη κυρία Χένκολα, αλλά έχετε ξεπεράσει τα τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σμόκρας. Πολλά ε, ενδιαφέροντα ερώτηματα έχουν τεθεί. Ένα ερώτημα έχω κι εγώ για την ε, μελέτη που έχετε κάνει. Είναι σωστό ότι στην ε, μελέτη που βλέπουμε για, την, για τις εκπομπές του γύρω 5 και γύρω 6 υπάρχουν λάθη στα δεδομένα και στην επεξεργασία τους, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι η αξιολόγηση θα είναι χωρίς λάθη ή έχουν υπάρξει όντω λάθη στην αξιολόγηση και θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Γιατί μιλάμε για μετρήσεις και για ακρίβεια. Πώς έγινε αυτό εσωτερικά, μπορείτε να μας ε, εξηγήσετε την ε, διαδικασία που ακολουθήσατε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πολύ καλή ερώτηση και συμπληρώνει και τις ερωτήσεις των προηγούμενων μελών. Βεβαίως πάντα γνωρίζουμε το θέμα της ε, ακρίβειας των μετρήσεων. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Δεδομένου και του ότι ελέγχουμε σε συνθήκες ε, κίνησης, ε, πάντα υπάρχουν ε, δυνατότητες, οι πιθανότητες να γίνουν λάθη, πάντα το ελέγχουμε αυτό, αλλά ένας τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι δεν αρχίσουμε να λέμε ότι τα δεδομένα μας είναι λάθος, είναι ότι, και το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, συζητούμε τα αποτελέσματα με τους εισαγωγείς, ανά αυτοκίνητο, τα δεδομένα δηλαδή του κάθε, του κάθε οχήματος, μετά τα αποτελέσματα που έχουμε, συζητούμε τα, μετά την, τη δοκιμή συζητούμε τα αποτελέσματα με τον, εισαγωγό και με τον εισαγωγέα και τον κατασκευαστή στις κατοχώρες. Οπότε υπάρχει έτσι μια ισορροπία στην διαδικασία γιατί και ο κατασκευαστή μπορεί να σχολιάσει τα αποτελέσματα. Ένα κομμάτι τη συζήτηση λοιπόν είναι ότι αν ένα όχημα, αν ένα όχημα είτε είναι στη σωστή λειτουργική κατάσταση, μπορεί κάποιο να πάει πίσω στον, στο εργοστάσιο και να δει αν έχουν υπάρξει προβλήματα συντήρηση. Αν υπάρχουν προβλήματα συντήρηση, τα λύνουμε και ξανακάνουμε τη δοκιμή. Οπότε υπάρχουν κάποιοι τέτοιε δικλείδε ασφαλεία και έχουμε και, την, ε, και ε, τον εξοπλισμό PEMS, ε, το οποίο εγκαθίσταται στο αυτοκίνητο και το όχημα βγαίνει σε συνθήκες κυκλοφορίας να δοκιμαστεί. Και στις δοκιμές που κάνουμε στα στα εργαστήρια, ελέγχουμε όλους τους αισθητήρες κτλ. Έχουμε, όπως είπα, και τους συντελεστές 3, 4, 5, 6 για τις εκπομπές που σημαίνει ότι εκπίπτει αυτό τη οποιασδήποτε συζήτηση για ακρίβεια. Γιατί αν είσαι 10%-20% εκτό των αποδεκτών ορίων, πάλι έχουν κάποια αξία τα αποτελέσματα αυτά, αλλά Άλλο ένα πείραμα που κάναμε και ήταν χρήσιμο για μας ήταν στην Σουηδία. Έγινε ε, έλεγχος με συστήματα στο πλάι του δρόμου ε, και από απόσταση και επιβεβαιώθηκε όντω ότι υπάρχουν υψηλέ εκπομπέ από τα οχήματα. Υπάρχει λοιπόν ε, και άλλη μέθοδο που επιβεβαιώνει και καταλήγει στα ίδια, σημεία, στα ίδια στοιχεία που καταλήξαμε κι εμεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τρέχουσα διαδικασία πόσο ακριβής είναι για να μετρήσει τα οξύδια του αζότου αν παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις διαφορές που υπάρχουν και εντός του εργαστηρίου και στις πραγματικές συνθήκες και με το συνδυασμό των διαφόρων παραγόντων για την, που θα μπορούσαν ίσως να επηρεάζουν την ανταλλαγή εκπομπών. Πόσο ακριβές είναι το σύστημα αυτό. Υπάρχει κάποια έρευνα σχετικά που να το υποστηρίζει. έγιναν κάποιες ε, ε, δοκιμές με τις ίδιες συνθήκες που υπάρχουν όταν γίνονται και τεστ, όταν γίνονται και δοκιμές. Δεν είναι το σαφέ σε τι ακριβώς αναφέρεστε, στις εγκρίσεις τύπου, σε άλλες δοκιμές. Η αξιολόγηση της ε, ακρίβειας είναι ένα κομμάτι της όλης διαδικασίας που γίνεται. Θα μπορούσαμε βεβαίω να σας ε, στείλουμε ίσω κάποιε γραπτές πληροφορίες. Ε, δεν τα ξέρω απ' τα στοιχεία. Είναι δυνατόν όμω να δω αν υπάρχουν τέτοιες, ε, τέτοια έγγραφα και να, αν είναι προσβάσιμα να σα τα αποστείλουμε. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που είστε εδώ, κύριε Σμόκερς. Έχετε κάποια εμπειρία δημιουργίας αυτών των ε, δοκιμών RDE και πόσος χρόνος χρειάζεται κατά την εμπειρία σας να δημιουργηθεί εξ αρχής ένα, μια τέτοια δοκιμή RDE. Ε, μπερδεύτηκα λίγο. Τώρα εκπονείται το RD, η δοκιμή των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Συγγνώμη, ε, όταν έχετε δημιουργήσει το σύστημα δοκιμής, είναι σύστημα εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες. Πόσο καιρό σας πήρε για να το εκπονήσετε αυτό το σύστημα. Α, μάλιστα εφαρμογή του RD, δηλαδή στο δικό μας πρωτόκολλο δοκιμών. Ε, έχουμε αρκετό καιρό που κάνουμε συζητήσεις και μάλιστα μας πήρε αρκετό καιρό μέχρι να ορίσουμε τις πρώτες λεπτομέρειες. Μόλις έγινε αυτό, μπορέσαμε να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες μέτρησης για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις, ε, τις εκπομπές σε συνθήκες πραγματικές. Πρόσφατα μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το σύστημα, ε, προσαρμόζουμε το πρόγραμμά μας λοιπόν μετρήσεων για να ε, συμπεριλαμβάνει και στοιχεία που είναι συμβατά με τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες. Οπότε πραγματικά μας παίρνει αρκετό χρόνο, γιατί ούτως ή άλλως και οι κατασκευαστές πρέπει να δαπανίσουν χρόνο σχετικά. Όλοι ούτε ή άλλως ε, σχεδιάζουν τα δικά τους συστήματα δοκιμών. Δεν είναι όμως κάτι που παίρνει χρόνια, ε, κάποιες εβδομάδες παίρνει για να δούμε, να δοκιμάσουμε το σύστημα για να δούμε ότι όντως ε, πληρεί τις προϋποθέσεις. Οπότε, αν κάποιος υπάλληλος σας δηλαδή έρθει και σας πει ότι θα πάρει δύο χρόνια θα τον απολύσετε, ε, θα πρέπει να του μιλήσω σίγουρα πριν τον απολύσω. κύριος σε λόγο. Ευχαριστώ. Να επανέλθω σε αυτό που απαντήσατε στην ε, ερώτηση 10 στο ΠΕΜΣ για το φορητό σύστημα ε, υπολογισμού εκπομπών. Είπατε ότι είναι 30%. Πολύ χαμηλό δεν είναι αυτό. Αν σε σχέση με αυτό που, αν μάλλον λάβουμε υπόψη αυτό που είπατε ότι ε, πιο πριν, ότι χρειάζεται μια δοκιμή για να μα αποδείξει ότι όντω γίνεται αυτό. Δηλαδή ζητούμε το, από τον κατασκευαστή να, το κάνει, να κάνει τη δοκιμή στο εργαστήριο, το κάνει στο εργαστήριο. Αν του πούμε να την κάνει σε πραγματικέ συνθήκε, την κάνει σε πραγματικέ συνθήκε. Αλλά πώ μπορούμε εμεί να κάνουμε τη μέτρηση. Είναι εφικτό να γίνει κάτι σε, ένα χρονικό, σε αυτό το χρονικό περιθώριο που, που συζητάμε, να το έχουμε δηλαδή, να έχουμε ένα λειτουργόν σύστημα το συντομότερο δυνατόν. Σε σχέση με την προηγούμενη απάντησή μου, η σκοπιμότητα του να γίνει η δοκιμή είναι ακριβώ για να μην υπάρχουν προβλήματα. Και η βασική ανησυχία του κατασκευαστή είναι να προσαρμόσει τα μοντέλα των οχημάτων έγκαιρα για να μπορεί να έχει διαφορετική απόδοση το όχημά του από ό,τι έχει τώρα. Και αυτό βεβαίω παίρνει κάποιο χρόνο και όταν έχει πολλά μοντέλα παίρνει περισσότερο χρόνο. Αυτή ίσω να είναι η μεγαλύτερη ανησυχία, αλλά το να γίνει, να είναι λειτουργών το σύστημα των δοκιμών δεν είναι, δεν είναι προβληματικό. Ναι, αλλά η γενική αξιοπιστία του συστήματος είναι 30% μας είπατε. Αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Εντάξει, για τους ε, κατασκευαστές είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά εμείς που θα νομοθετήσουμε. Πώς θα το δοκιμάσουμε με τόσο χαμηλή αξιοπιστία, πώς θα βασιστούμε σε αυτό για να νομοθετήσουμε. Ε, εντάξει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το αξιολογήσετε. Για τα roller banks υπάρχουν ε, αρκετά στοιχεία που σημαίνει ότι πρέπει στην νομοθεσία σας να έχετε διατάξεις που ασχολούνται σχετικά. Αν δηλαδή η πρώτη δοκιμή δεν είναι συμμορφούμενη, την ξανακάνετε. Υπάρχουν διαδικασίες για το πόσα τις δοκιμές μπορείτε να κάνετε πριν εξασφαλίσετε ότι τα στατιστικά σας είναι επαρκώς αξιόπιστα για να πείτε ότι να είμαστε πάνω από το όριο. Τώρα, αν η μέθοδος υπολογισμού είναι ανακριβής, τότε πρέπει να έχετε πολύ περισσότερα στατιστικά πριν καταλήξετε σε ένα αποτέλεσμα που να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τις διατάξεις και το χρονικό όριο που βάζετε μέσα στην νομοθεσία σας για να γίνει αυτό. Υπάρχουν τα, η έγκριση τύπου για τα roller banks. Υπάρχουν διαδικασίες που, μπορεί να σας, μπορούν να σας βοηθήσουν να περιγράψετε ποιο είναι το follow-up, η παρακολούθηση. Και αυτό μπορεί να γίνει παρόλο που χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια γιατί δεν είναι τόσο παρκές. Δηλαδή όταν κάποιος ε, έχει κακό αποτέλεσμα στην δοκιμή, το ξανακάνει και το ξανακάνει από την αρχή. Αυτό λέτε. Ε, δεν θα ήθελα τώρα να μιλάμε για άσχημα αποτελέσματα, ας πούμε, έλα, ε, όχι αρκετά αξιόπιστα. Ναι, ευχαριστώ. Για να είναι λίγο σαφή τα πράγματα, γιατί είπατε αρκετές φορές ότι δεν είναι δεν είστε σίγουρος ότι μπορεί κανείς να επιτύχει τους στόχους στην πραγματική χρήση. Αλλά στην απάντησή σας στην ερώτηση 1 λέτε σαφές ότι καμία νέα τεχνολογία δεν χρειάζεται για να επιτύχουμε χαμηλότερες εκπομπές οξυδίου του αζότου στις πραγματικές συνθήκες. Αυτό τι σημαίνει, ότι με τις τρέχουσες τεχνικές θεωρείτε ότι μπορούμε να επιτύχουμε τα τρέχοντα πρότυπα που έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 80 μιλιγκράμμ δηλαδή ανά χιλιόμετρο. Αυτό ακριβώς λέμε με βάση την αξιολόγηση των εμπειρογνωμών μας. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες, σχεδιάζονται τώρα σε συγκεκριμένα ε, στοιχεία για, το, αν για να δούμε αν εφαρμοστούν στον κινητήρα μπορούν να λύσουν το πρόβλημα ή όχι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει έτσι μια ε, κλιμάκωση στο σύστημα, να δούμε αν ε, υπάρχει δυνατότητα ελέγχου που να μπορεί να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα σε συνθήκες πραγματικές. Ναι, αλλά αν δούμε τις διαφορετικές τεχνικές που υπάρχουν, είσαστε αρκετά επικριτικός ε, για το EGR συγκεκριμένα. Έτσι δεν είναι. Ουσιαστικά δεν θεωρούμε ότι το Euro 6 μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το EGR. Πρέπει να υπάρχει EGR με LNT ή EGR με SCR. Συνδυασμός. Από μόνο του δεν ε, αρκεί. Το εξηγώ και στο κείμενο. Και αυτό είναι ευρέως γνωστό. Θεωρούμε πως ναι. Άρα αν τα νέα, τα οχήματα που ε, τίθενται σε εμπορία στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν μόνο στη τεχνολογία EGR θα σας σόκαρε. Αν ε, είναι πιο καθαρά και μπορούν να πληρούν τις προποθέσεις για τις διάφορες συνθήκες, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και δυνατό αυτό που λέτε. Άρα θα έχουμε ε, ερώτηση προς την αυτοκινητοβιομηχανία αν, παρέ, αν παράσχει μόνο αυτοκίνητα στην αγορά που έχουν συν, τεχνολογία EGR. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, κύριο Σμόκερς και τον κύριο Κίλνερ για την παρουσία τους, για την υπερογνωμοσύνη τους. Ξέρω ότι δεν μπορέσατε να απαντήσετε σε όλα τα ε, ερωτήματα. Κάποια ήταν πολιτικής φύσεως, κάποια νομικής. Αλλά θα ήθελα να πω στους συναδέλφους μην ανησυχείτε, θα επανέλθουμε στο θέμα. Ίσως οι συνάδελφοι να έχουν και κάποιες τεχνικές ερωτήσεις, τις οποίες θα σας στείλουμε βεβαίως ε, και ελπίζουμε ότι θα μας απαντήσετε και σε αυτές. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Um, Συνάδελφοι, να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της ε, ακροασής μας. Με δύο πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Πολύ γνωστό οργανισμό σε όλους μας, σε όποια επιτροπή και αν συμμετέχουμε, ΔΕΒΕ, ΙΝΤΑ, να καλωσορίσω τον ε, κύριο Πολ Μακάλαβη που είναι επικεφαλής του προγράμματος ε, για την κλιματική αλλαγή και τον κύριο Μάρτιν Άνταμς που είναι επικεφαλής της ομάδας ε, ρήπανσης του αέρα, μεταφορών και θορύβου. Κύριε Μακάλαβη, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή σας που μας απίφευε την πρόσκληση. Εγώ και ο Μάρτιν θα σας παρουσιάσουμε κάποιες διαφάνειες και στην εισαγωγική μας παρουσίαση θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όσον αφορά την εντολή του οργανισμού μας θα πούμε δύο λόγια για τις ε, δραστηριότητες μας, για τα οξύρια του Αζίτ, για την κατάσταση της ποιότητας του αέρα και πώς αυτή συνδέεται με τις εκπομπές και τέλος θα μιλήσουμε για το πώς ο οργανισμός μας ε, κοινοποίησε τις γνώσεις και τις, και τις πληροφορίες που συνέλεγε για τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες την τελευταία δεκαετία. Εντολή του EEA, η εντολή αυτή έχει οριστεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και αναφέρεται ρητός ότι πρόκειται για έναν φορέα παροχής γνώσεων. Δεν μας έχει ανατεθεί ρόλος στην δοκιμή ή στην μέτρηση, ούτε έχουμε εξουσίες ε, ελέγχου και επιθεώρησης. Ωστόσο, η εντολή μας μας παρέχει έναν σημαντικό ρόλο προκειμένου να παρέχουμε στην κοινότητα και στα κράτη-μέλη αντικειμενικές αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου εκείνοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος να αξιολογούν τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων και να εξασφαλίζουν ότι η δημόσια, ε, το, το κοινό ενημερώνεται με τον κατάλληλο τρόπο για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Εμείς επίσης συντάσσουμε μια ετήσια έκθεση για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ε, με βάση στοιχεία που μας παρέχουν αυτοκινητοβιομηχανίες και κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τον ε, κανονισμό ε, συντάσσουμε και την ετήσια έκθεση για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πάλι στη βάση των υπολογισμών των κροτών μελών. Ε, οι δικές σας ερωτήσεις αφορούν περισσότερο τους ρυπογόνους παράγοντες του αέρα. Να σας πω ότι εμείς ε, ε, ασχολούμαστε και με το θέμα των πραγματικών εκπομπών οξυδίων του αζότου. Επίσης, εδώ μπορείτε να δείτε και το θέμα του κόπερτ Βοηθούμε τα κράτη-μέλη στην ε, σύνταξη και στη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών. Θα σας πει κάποια λόγια περισσότερα για αυτό το θέμα και ο Μάρτιν. Επίσης υποβάλλουμε έκθεση για τα δεδομένα παρακολούθησης ποιότητας αέρα που μας υποβάλλουν τα κράτη-μέλη στη βάση των δικών τους ε, μετρήσεων για το διοξίδιο του αζότου. Ο Μάρτιν θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα ευρήματά μας σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Όπως περιγράφηκε, ο οργανισμός ασχολείται με διάφορα τύπη, διάφορους τύπους ε, εκπομπών ε, και οχημάτων. Τα νέα επιβατικά οχήματα είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, ο σύνολο τουλάχιστον, έχει ήδη ε, επιτύχει τον στόχο του 2015 για 130 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρα. Ωστόσο, οι ε, μετρήσεις, οι εργαστηριακές, είναι χαμηλότερες από αυτές που υπάρχουν σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης βλέπουμε από τα επίσημα στοιχεία που μας υποβάλλουν τα κράτη-μέλη ότι ε, οι επιδόσεις του κλάδου δεν είναι πολύ θετικές. Αντιθέτως, σε σύγκριση με το 1990, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί κατά 17%. Και μάλιστα είναι ο μόνος κλάδος ε, της οικονομίας στην, οι, οι, οδικές μεταφορές ε, στον οποίο οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί. Πραγματικές εκπομπές NOx εδώ έχουν μειωθεί σημαντικά κατά σχεδόν 60% 100, τα τελευταία 25 χρόνια. Ωστόσο, είναι σαφής, σαφές ότι η μείωση αυτή θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν τα τζελοκίνητα οχήματα είχαν ανταποκριθεί στα πρότυπα Euro. Όπως έχει συμβεί με τα πετρελαιοκίνητα. Ο χάρτης αυτός αποτυπώνει ε, την, ε, τις μετρήσεις διοξιδίων του αζότου, όπως μας υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Βλέπετε εδώ ότι οι κόκκινες ε, βουλίτσες ε, είναι τα κέντρα ελέγχου και δοκιμών. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια κέντρα σε πολλές χώρες. Βλέπετε ωστόσο ότι σε πολλές ε, περιφέρειες και σε πολλές περιοχές υπάρχει ε, υπέρβαση των επιτρεπόμενων όριων. 19 συγκεκριμένα. Στις περιοχές όπου υπάρχει ε, υπέρβαση, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της υπέρβασης οφείλεται στις οδικές μεταφορές. Για μας αυτό είναι σημαντικό ε, λόγω του κινδύνου και της βλάβης που προκαλούν τα, τα οξύδια του αζότου στην ε, υγεία του ανθρώπου. Μαζί με τα ε, μικροσωματίδια, ε, τα οξύδια του αζότου είναι από τους πιο επικίνδυνους ρυπογόνους παράγοντες. Κόπερτ. Ε, μας υποβάλλατε και κάποιες ερωτήσεις για αυτά τα θέματα. Θα σας εξηγήσω λίγο τι ακριβώς είναι το Copert. Το Copert λοιπόν είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη, σε επιστήμονες, ερευνητές να εκτιμούν ποιες είναι οι πραγματικές εκπομπές του κλάδου των μεταφορών. Τόσο για τα οξύδια του αζότου, όσο και για το διοξείδιο του άνθρακα και άλλους ρηπογόνους παράγοντες ως ε, οργανισμός έχουμε υποστηρίξει την ανάπτυξη αυτού του software για πάνω από μια δεκαετία σε συνεργασία και με το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Κομισιόν. Και σκοπός είναι να ε, παρέχονται αξιολογήσεις για τις πραγματικές εκπομπές με βάση τις, ε, τα, τις επιστημονικές ενδείξεις που έχουμε από ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η τελευταία μας διαφάνεια όπου και προσπαθούμε να ε, συνοψίσουμε τις δημοσιεύσεις που έχει κάνει ο οργανισμός μας τα τελευταία χρόνια. Ε, μία από τις, τις ερωτήσεις σας ήταν αν πότε ε, η, ο EEA διαπίστωσε αυτή αυτό το χάσμα μεταξύ των πραγματικών και των εργαστηριακών μετρήσεων. Εμείς εξετάσαμε όλες τις εκθέσεις που είχαμε υποβάλει και δημοσιεύσει τα τελευταία 10 χρόνια για να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί και διαπιστώνουμε από το 2004 φαινόταν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ε, οι μετρήσεις ε, στα εργαστήρια δεν αποτύπωναν με μεγάλη ή με απόλυτη ακρίβεια τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες. Ε, και αυτό βασίστηκε σε γνώσεις που συλλέγαμε ε, στο θέμα της ποιότητας του αέρα. Τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερο είχαμε ενδείξεις για αυτήν την απόκληση και το 2010 ε, και 2010 στις ε, εκθέσεις μας για το ευρωπαϊκό περιβάλλον θέσαμε αυτά τα θέματα. Πέρσι ε, αποφασίσαμε μάλιστα να εκδώσουμε ένα εγχειρίδιο για να εξηγήσουμε τις ε, οδηγίες και τις συστάσεις μας ε, ε, στο ευρύ κοινό. Το κάναμε αυτό μάλιστα πριν και από τις αποκαλύψεις του τελευταίου Σεπτεμβρίου για τις, συσκευές, για τις διατάξεις Στο ερώτημά σας, αν θα έπρεπε οι υπερβάσεις αυτές να είχαν εντοπιστεί από κάποιον ευρωπαϊκό οργανισμό νωρίτερα, εμείς μπορούμε να σας απαντήσουμε ότι το 2004 είχαμε εντοπίσει αυτό το στοιχείο αλλά, ε, και το είχαμε δημοσιεύσει, αλλά βεβαίως δεν είμαστε η μοναδική φωνή. Επειδή ακριβώς είμαστε φορέας παροχής πληροφοριών, εμείς θα ε, αντλούμε μάλλον το δίδαγμα από την ιστορία αυτή ότι θα πρέπει να κατευθύνουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις ε, πληροφορίες και τις γνώσεις που συλλέγουμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η, η συμβολή μας είναι θετική τόσο όσον αφορά την, ε, την ποιότητα του αέρα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση και την, προστασία της βιοπικιλότητας. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, ε, θέλουμε να σας πούμε ότι σας, εκτιμούμε, ότι σας εκτιμούμε εσάς και τις εργασίες της Επιτροπής σας πάρα πολύ και βεβαίως δεσμευόμαστε ότι αν υπάρξουν ερωτήσεις σήμερα τις οποίες δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε γραπτό στις απαντήσεις μας ε, μετά τη σημερινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ ε, να περάσω στους συγητές μας, ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακαλίβη και κύριε Άνταμς για την παρουσία σας εδώ. Λέτε ότι προειδοποιούσατε τους φορείς χάραξης πολιτικής από το 2004 για το χάσμα μεταξύ εργατιστηριακών και πραγματικών μετρήσεων. Και μάλιστα ανησυχείτε και για τις επιπτώσεις που έχει αυτό το χάσμα στην ε, ποιότητα του αέρα και ότι δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχουμε τους στόχους μας αν το χάσμα αυτό διατηρηθεί. Ε, προφανώς ε, εσάς δεν σας ενδιαφέρει το πώς τα αυτοκίνητα θα μπορέσουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Αλλά γνωρίζω τον οργανισμό σας πολύ καλά και ξέρω ότι συμμετέχετε σε πολύ δραστήρια στις συζητήσεις μεταξύ του JRC, της Κομισιόν, αλλά παρίσταστε και σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν ε, λίγα περισσότερα πράγματα για το τι είδους απαντήσεις λαμβάνατε από το 2004 όταν και αρχίσατε να προειδοποιείτε τους, φορείς, ε, τους διάφορους φορείς. Ποιες ήταν οι απαντήσεις που σας έδιναν στις προειδοποιήσεις σας αυτές το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξαμε το χρονοδιάγραμμα των εκθέσεων της τελευταίας δεκαετίας και πόσες φορές, φορές ε, επισημάναμε αυτό το θέμα. 28 σε 12 χρόνια. 28 φορές θέσαμε το θέμα της απόκλησης μεταξύ εργαστηριακών και πραγματικών ε, μετρήσεων. Εμείς βασιστήκαμε σε δεδομένα οργανώσεων όπως το TNO ε, από το 2011 και 2010-2011 και έπειτα όλο και πιο συστηματικά Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτική θα πρέπει να χαράσετε με βάση στοιχεία και ενδείξεις πραγματικές. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε η μοναδική φωνή στις συζητήσεις αυτές. Από το 2010-11 και έπειτα, και ομολογώ ότι ήταν η προκάτοχή μου, όχι εγώ, σε αυτές τις συζητήσεις, που ιδίω οι συνάδελφοι της ε, Γενικής Διεύθυνση Περιβάλλοντος συνειδητοποιούσαν την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτή η απόκληση και συζητούσαν έντονα το θέμα αυτό και στο διεθνές πλαίσιο, στο πλαίσιο του UNEC, τα κράτη-μέλη συζητούσαν αυτό το θέμα και είχαν επίγνωση της δυσκολίας επίτευξης α, αυτού του στόχου περί του χάσματος. Ναι, είπατε 2010-2011 ότι από την DG Envy είχατε λάβει κάποιες απαντήσεις στις εκθέσεις που υποβάλατε εσείς. Εσείς αντιληφθήκατε να υπάρχουν τίποτα εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ DG Envy και Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας. Ε, αυτά τα θέματα συζητήθηκαν εσωτερικά στην Κομισιόν. Έχετε κάποια τέτοια εικόνα. Επίσης, συζητήσατε όλα αυτά τα θέματα με τους συναδέλφους σας από το Κοινό Κέντρο Έρευνας. Ο Πολ είπε για, το 2000, για τα στοιχεία του 2004. Το 2007 ήδη είχαμε διοργανώσει κάποια σεμινάρια, κάποια εργαστήρια ε, σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Έρευνας για την απόκληση. Ε, το 2010 η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος είχε διοργανώσει επίσης μια διαβούλευση με εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη ε, με στόχο, με θέμα μάλλον, τις αποκλίσεις που υπήρχαν μεταξύ πραγματικών και εργαστηριακών μετρήσεων. Ε, εμείς, ο βασικός μας ε, εταίρος είναι η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Και δεν σας είπε κανείς έστω και ανεπίσημα ότι δέχονται πιέσεις από την Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας. Όχι, λέει ο, ο μιλητής, δεν σας πιστεύω, λέει ο κύριος Βουλευτής. θα ήθελα να μου πείτε αν βλέπετε να υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και αν ε, υπάρχουν τέτοιου είδους αδυναμίες ε, πώς εκφράστηκαν πρακτικά. Μιλώ πάντα για τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Οι σχέσεις μας με τα κράτη-μέλη είναι ποικίλε. Είναι και αυτές που είπατε εσείς, αλλά και οι τεχνικές συναντήσεις που διοργανώνουμε ε, για την κατάρτιση των επίσημων εκθέσεων για τα NOX. Υπάρχουν ε, επίσημες κοινότητες εμπειρογνωμόνων όπου και συζητούμε αυτά τα, ζητήματα. Το Κόπερτ είναι ένα παράδειγμα. Επίσης, στόχος της, του οργανισμού μας είναι να δίνουμε καθοδήγηση προς τα κράτη-μέλη για το πώς μπορούν να εκτιμούν ή να μετρούν τις ε, εκπομπές τους. Ε, εκδίδουμε και ένα σχετικό εγχειρίδιο με μεθοδολογίες ε, τις οποίες μπορούν να εφαρμόζουν ε, οι εθνικές αρχές. Θεωρείτε ότι υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά την συνεργασία σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπαμε, η συνεργασία μας με την Κομισιόν είναι πάρα πολύ στενή. Εμείς ως οργανισμός δεν ξέρω αν το ξέρει η Επιτροπή σας, ε, ο οργανισμός μας λοιπόν έχει ένα διοικητικό συμβούλιο όπου εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη με ένα μέλος και η Κομισιόν με δύο μέλη. Υπάρχει και ένας εμπειρογνώμονος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα το βασικό, ο βασικός διάβλος επικοινωνίας μας με την Κομισιόν είναι αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την τεχνική συνεργασία, αυτή αφορά πάντα τις πραγματικές εκπομπές, την ποιότητα του αέρα και όπως είπε και ο κ. Γκυρμπράντη υπάρχει μια μακρά και στενή συνεργασία με τους συναδέλφους από τη Eurostat, από το JRC, την ε, Γενική Διεύθυνση Κλιματικής Δράσης, την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Συνεργαζόμαστε και με τη Γενική Διεύθυνση MOVE. Όλο και, περισσότερες, όλο και στενότερη συνεργασία μας με, είναι με την Digimare και έχουμε την αίσθηση ότι η συνεργασία μας είναι αποτελεσματική. Για το ερωτηματολόγιο να σας ρωτήσω κάτι. Στην ε, σελίδα 8 των απαντήσεών σας είπατε ότι ε, ε, τα μικροσωματίδια έχουν μειωθεί κατά 50% σε σύγκριση με το 1990. ενώ οι εκπομπές από τα υδραυλικά φρένα έχουν αυξηθεί. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Ναι, είναι πρόβλημα. Το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Η αποδοτικότητα των ε, σωματιδιακών φίλτρων έχει ε, βελτιωθεί σημαντικότητα και ως εκ τούτου τα ε, σωματίδια που εκπέμπονται από τους νέους κινητήρες είναι πολύ πολύ λιγότερα. Πάντως εμείς σε κάθε περίπτωση βασιζόμαστε στις εκτιμήσεις και στις μετρήσεις των κρατών μελών. Σε απόλυτους αριθμούς ε, τα σωματίδια έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί οι μεταφορές, περισσότερα οχήματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Έρευνας που ε, θα μπορούσε ή που αυτό τον καιρό ε, ασχολείται με, την, με τον εντοπισμό συγκεκριμένων ε, πηγών για, αυτές, για αυτά τα σωματίδια. Κύριος Κάρετς. Μου θυμίζει η σημερινή συνεδρίαση με, το JRC, με τη, τη που είχαμε με το JRC. Εσείς, αφού είχατε εντοπίσει το πρόβλημα το 2014, ε, το 2004, συγγνώμη. Έχουν περάσει 12 χρόνια. Έχουμε 2016. Πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει νομοθετικά. Οπότε εγώ συμπεραίνω ότι σίγουρα υπάρχουν υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που σας έχουν πει Παιδιά κάντε στην πάντα, μην τα βγάζετε στην ε, δημοσιότητα αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να μου πείτε ποιοι ήταν αυτοί, αυτά τα πρόσωπα. Εγώ προσωπικά ε, δεν έχω επαφές με επικεφαλής ε, κυβερνήσεων και κρατών. Όχι, εντάξει, ας σοβαρευτώ. Από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος δεν έχουμε καμία πληροφορία η οποία μας απαγορεύτηκε να τη δημοσιεύσουμε ή που σκοπίμως δεν δημοσιεύσαμε. Όχι, καταλαβαίνω ότι δημοσιεύσατε, αλλά ε, ε λέτε δηλαδή ότι δεν, δεν έχει υπάρξει ούτε ένας πολιτικός ο οποίος να προσπάθησε να σας εμποδίσει στο έργο σας. Ό,τι κάνατε, το κάνατε πλήρως ανεμπόδιστα, με κάθε ελευθερία. Όχι. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Κανένας πολιτικός δεν έχει προσπαθήσει να σταματήσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος από το να δημοσιεύει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του. Ωραία. Αν δεν υπήρξε κανένας πολιτικός που να το έκανε αυτό, τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να αλλάξουμε στο σύστημα. Γιατί με εκπλήσει. Λέτε ότι έχετε ε, καταπληκτική συνεργασία με τις γενικές διευθύνσει και παρόλα αυτά φτάσαμε στην κατάσταση στην οποία φτάσαμε. Ε, ε εσείς τι θέλετε να γίνετε, να, να γίνετε ένας υπεροργανισμός με εκτελεστικές εξουσίες. Ε, γιατί συγγνώμη, αν δεν σας εμπόδισε κάποιος πολιτικός να δημοσιεύσετε τις πληροφορίες αυτές, τότε μάλλον το σύστημα είναι χάλια να σας πω. Έχω μπροστά μου ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο, ε, ε, ε, εσωτερικό δικό μας, συγγνώμη, το οποίο έχουμε παρουσιάσει εδώ στο Κοινοβούλιο 10 Νοεμβρίου 2011 όταν ήρθαμε στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ερχόμαστε κάθε χρόνο και παρουσιάζουμε την σχετική έκθεσή μας για τις μεταφορές και εκεί ε, παρουσιάσαμε λοιπόν την έκθεση για το 2011. Φοβόμασταν ενδεχομένως ότι ήταν πάρα πολύ εκτενής η έκθεση και έτσι είχαμε συντάξει μια δισέλιδη ε, σύνοψη την οποία και διαβάσαμε εδώ όπου ήταν πάρα πολύ σαφές όπως, όπως είπα 10 Νοεμβρίου 2011 και εκεί λέγαμε συνολικά οι στόχοι υπερβαίνονται σε πάρα πολλούς τομείς υπάρχει, πρέπει να εξηγηθούν οι ε, διαφορές μεταξύ των εκπομπών και των ε, στόχων ε, για την ποιότητα του, ε, του αέρα. Υπάρχει μεγάλη διάδοση των ε, διζελοκίνητων οχημάτων και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πραγματικές εκπομπές των οχημάτων είναι μεγαλύτερες από τις εργαστηριακές. Το είπαμε στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, εντάξει, ε, ίσως θα έπρεπε να είχαμε, ε, να είχαμε επιμείνει περισσότερο. Και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Μεταφορών τι σας είπαν, πηγαίνετε στο διάολο ή είπαν ότι θα κάνουμε κάτι με αυτά τα στοιχεία που μας φέρνετε. Εσείς απλά διαβιβάσατε αυτές τις πληροφορίες. Ε, τι, τι, τι ακριβώς κάνατε δηλαδή. Ε, ναι, είναι μία παράγραφος αυτή. Ναι, η οποία είναι κρυμμένη μέσα σε μια δισέλιδη ε, σύνοψη. Ε, different MEPs reacted in different ways διάφοροι ευρωβουλευτές είχαν διάφορες αντιδράσεις. Τι θέλετε να σας πω τώρα. Υπάρχει κάποιο μέλος της Επιτροπής Μεταφορών. Η κυρία Μπονεφουά. Je voulais poser un peu la même question. Je vais vous la reposer pour plus précisément vous indiquer. Μπορείτε να μας πείτε το 2011 ήρθατε ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών για να δώσετε τις πληροφορίες. Χρειάστηκε να περιμένουμε η Δανέζα υπουργό Περιβάλλοντος να στείλει επιστολή το 2013 για να επιταχυνθούν τα πράγματα. Ή διάβασα τις απαντήσεις που δώσατε στην πρώτη ερώτηση για να εξηγήσετε την αυστηρή σας εντολή και ότι δεν μπορείτε να την ξεπεράσετε και ότι στις απαντήσεις στη 4 όσον αφορά τις ομοσπονδιακές, τους ομοσπονδιακούς οργανισμούς της Αμερικής Βλέπουμε τη διαφορά. Γιατί εκεί έχουν πολύ περισσότερο προσωπικό και τη δυνατότητα να ελέγξουν τις ε, ρυθμιστικές διατάξεις και να υποβάλουν και προτάσεις. Ξέρω πως δεν είναι αυτή η εντολή σας σήμερα. Αλλά όπως είπε ο συνάδελφος και πριν, πρέπει εμείς να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Εσείς τι θα προτείνατε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ως εντολή για να είστε πιο αποτελεσματικοί και πέρα από την επικοινωνία να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή των κανόνων και ε, στην, ε, στον περιορισμό των εκπομπών ρήπων. Thank you uh, for the question. Um, it's... Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, γι' αυτό ξεκίνησαμε αυστηρές τι εξηγήσει. Είναι σαφέ ότι ο έλεγχο τη συμμόρφωση δεν είναι κομμάτι τη δική μα εντολή, δεν έχει συζητηθεί στο Διοικητικό μα Συμβούλιο και τελικά, όπω είπατε, αν υπάρχει μια αλλαγή στην εντολή τη υπηρεσία, αυτό είναι θέμα των ε, θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών να το κάνουν. Αν εσεί θεωρείτε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντο να έχει στις αρμοδιότητες της και τον έλεγχο της ε, συμμόρφωσης θα είναι σημαντική θεμελιώδης αλλαγή των ε, εργασιών μας. Και θα έδινε διαφορετική έμφαση στη φύση της δουλειάς μας και θα εισήγεται έτσι και πρώτη φορά ο έλεγχος συμμόρφωση. Δεν είμαι σίγουρο κατά πόσο το Συμβούλιο θέλει κάτι τέτοιο, να έχει δηλαδή τέτοιε αρμοδιότητε η υπηρεσία περιβάλλοντος. Αυτή η συζήτηση δεν νομίζω ότι είναι επίκαιρη αυτή τη στιγμή. Τώρα, κατά δική μου την άποψη την προσωπική, θα ήταν απαραίτητο όποια αλλαγή γίνει στην έντολή μας να, να έχει και, τις και τους απαραίτητους πόρους και την απαραίτητη πολιτική ε, στήριξη. Γιατί αλλιώ δεν θα έχουμε απαραίτητα ε, τα, καλά, τα σωστά αποτελέσματα. Γιατί η φήμη μα τα τελευταία χρόνια βασίζεται στην ανεξαρτησία, στην αξιοπιστία. Και νομίζω ότι τον... Ε, δανείσουμε το όνομά μας σε ένα ε, αδύναμο νομισματικό σύστημα δεν είναι κάτι που θέλουμε κατά ανάγκη. Ε, σε σχέση με την ποιότητα του αέρα, ο οργανισμός μιλά στο τέλος για την αμμονία και το... και το υπεροξίδιο του αζότου οι τεχνολογίες κατά της ρήπανσης επιτρέπουν να περιοριστούν και να μην αυξηθούν στα επόμενα χρόνια. Και πρέπει να νομοθετήσουμε και για τις εκπομπές ε, αερίων. Και έπειτα μιλήσατε για τη θανατηφόρο επίπτωση του διοξιδίου του αζότου, αλλά όχι για το οξύδιο του αζότου. Ποιος είναι ο αριθμός των θανάτων, των αναπνευστικών ε, παθήσεων στην Ευρώπη σε σχέση με το οξύδιο του αζώτου και αν ο κανόνας 3-4 για τα ρούμενα σωματίδια είχε αρχίσει να ισχύει, πόσους θανάτους θα είχαμε μπορέσει να αποφύγουμε. Uh, starting with the final question about Euro 4 particulate matter, if that had uh, reached the necessary standards, what the impact would have been. Ποιο θα ήταν ο αντίκτυπο για του πρώιμου θανάτου αν είχε εφαρμοστεί νωρίτερα αυτό ο κανόνα. Δυστυχώ δεν έχουμε τέτοιε στατιστικέ. Ε, τώρα, για την αμμονία και το ε, υπεροξίδιο του αζότου. Η αμμονία βέβαια είναι παραπροϊόν στις τεχνολογίες ECR. Υπάρχει ίσως μια κάποια μικρή ανησυχία για υψηλά ποσοστά αμμονία σε κάποιες πόλεις. Το πρόβλημα με την αμμονία είναι ότι σχηματίζει σχηματίζει ε, ιδιαίτερες, ε, ιδιαίτερα συμπαγή σωματίδια που είναι ε, βλαβερά για το αναπνευστικό μας σύστημα. Τώρα, για το οξύδιο του αζότου και για τα μυρωμένα σωματίδια μπορούμε να τα ελέγξουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε μήπως τι γίνεται σε μη κανονικές συνθήκες, ώστε να βελ, βελτιστοποιηθεί το εξοπλισμός. Χένκελ. Yes, we <clears throat> Μας είπαν ότι ενημερώσατε την Επιτροπή και το κοινό σε 28 εκθέσεις στη διάρκεια 12 ετών και δεν έχει γίνει τίποτα. Ακούσαμε και διάφορες ερωτήσεις ε, και έφτασα στο συμπέρασμα ότι χωρίς τη ΣΥΠΑ και χωρίς το σκάνδαλο της Volkswagen, αυτό το θέμα δεν θα είχε συζητηθεί τόσο ευρέως όσο τώρα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό το συμπέρασμα it's, ναι, Από τον περασμένο Σεπτέμβριο και τις αποκαλύψεις για τις συσκευές αναστολής, ο αριθμός ετοιμάτων από, για να σχολιάσουμε αυτό το θέμα εμείς αυξήθηκε κατακόρυφα. Είπατε όμως ότι δεν συνέβη τίποτα με όλο το σεβασμό εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρχαν προτάσεις, αναπτύχθηκαν προτάσεις τα τελευταία χρόνια ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της απόκλησης. Ο χρονισμός είναι κάτι που εσείς ε, εξετάσατε όταν είχατε εδώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Απλά θα πρέπει να πω ότι δεν είναι ότι δεν συνέβη αποκλήτως, τίποτα. Ναι, το δέχομαι. Οπότε έγινε η δήλωση, μάλλον ε, τέθη το ερώτημα, κατά πόσο οι πολιτικοί ε, ενημερώθηκαν για αυτή τη γνωμοδότηση. Πολιτικοί ηθήνοντες. Βεβαίως, στείλατε την ε, έκθεση αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην Επιτροπή Μεταφορών. συμφωνείτε μαζί μου, ενημερώσατε καταλήλως το Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο το ίδιο όμως δεν ανέλαβε δράση. Δεν πρέπει σε ενέργειες. Ενέργειες που ζητάμε να αναλάβουν να κάνουν τώρα άλλη πολιτικοί. I, would, I would be to uh, εγώ δεν μπορώ να καταλήξω αυτό το συμπέρασμα, ότι δηλαδή το Κοινοβούλιο δεν ανέλαβε δράση. Εμάς μας ρωτήθηκε πότε γνωρίζαμε αυτού του είδους την απόκληση ανάμεσα στις ε, ε, εργαστηριακές ε, και στις πραγματικές συνθήκες. Εμείς όταν το αντιληφθήκαμε ενημερώσαμε τα κρατημέλη, ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα διαπιστώσαμε. Το θέμα της πενταετούς έκθεσης για το περιβάλλον είναι μια νομική υποχρέωση. Κάθε πέντε χρόνια να κάνουμε μια αναπογραφή για το ευρωπαϊκό περιβάλλον, καθώς και για τις προοπτικές του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Και αυτό το κάναμε. Τρεις τελευταίες για το 2005, 2010 και 2015. Και τα παρουσιάσαμε αυτά, τα υποβάλαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο. και αναφερθήκαμε στο θέμα της απόκλησης. Πιστεύουμε ότι εμείς πληρώσαμε την εντολή μας να προσφέρουμε πληροφορίες. Τελευταία μου ερώτηση. Πότε ακούσατε ότι οι κατασκευαστές μπορούν να χειραγωγήσουν τα αποτελέσματα μέσω software λογισμικού. Πότε το ξέρατε αυτό ότι γίνεται. Όταν ε, ε, θίξαμε το θέμα αρχικά το 2004, εμείς στηρίζαμε αυτό το μοντέλο και γιατί υπήρχαν όλα ένα και περισσότερες αποδείξεις ότι οι πραγματικές ε, εκπομπές δεν αντιστοιχούσαν στις εργαστηριακές. Τώρα κατά πόσο αυτό ρυθμιζόταν με software ή όχι, δεν το γνωρίζαμε. Πάντως, αυτοί οι λόγοι ήταν γνωστοί εδώ και αρκετό χρόνο. Πρώτον, κύκλος της δοκιμασίας. Δεύτερον, ευελιξία σε σχέση με το πρωτόκολλο των δοκιμών και έπειτα πραγματική συμπεριφορά οδήγηση, δηλαδή γρήγορε επιταχύσει, έντονε επιταχύσει κτλ. Υπήρχαν αυτοί οι τρει βασικοί λόγοι στου οποίου οφειλόταν οι διαφορέ και αποκλήσει. Τώρα, αν γινόταν χειραγώγηση και με λογισμικό, δεν το γνωρίζαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν σας βάλω στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Εσείς έχετε, έχετε απαντήσει ε, και τα σαφείς, προσπαθήσατε να γνωστοποιήσετε τα στοιχεία. Αυτό που μας μπορείτε να μας βοηθήσετε, δεν σας κατηγορώ, αλλά σε έναν κόσμο που θα είχατε εσείς λόγο. Βέβαια είναι πολιτική απόφαση, αλλά Πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει ότι τα απορίσματά σας θα διαβιβάζονται στο πολιτικό επίπεδο και θα τονίζονται. Γιατί εσεί είστε υπάλληλοι ενό οργανισμού. Δεν, δεν μπορείτε εσεί να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη. Εγώ όμω μπορώ να το κάνω, για απαντώντα ε, στον κύριο Χένκελ βεβαίω. η αντίδραση από την πλευρά του Κοινοβουλίου δεν ήταν επαρκή, αλλά αυτό είναι δικό μου ρόλο ως πολιτικού να το κάνω και να διαμαρτυρηθώ γι' αυτό. Αλλά αν υπήρχε ένα σύστημα όπου τα δικά σα πορίσματα θα μπορούσαν να τονιστούν και να είστε σίγουροι ότι διαβιβάζονται σε πολιτικό επίπεδο. Θα, πιστεύετε, πούμε, ότι θα έπρεπε να γίνονται αιτήσια ακροάσει ή ενημερωτικά έγγραφα. Ναι, ο κύριος Κάνε το είπε στην εισηγησή του ότι δεν τα διαβάζει κανεί. Ίσως κάποιος τρόπος να βρούμε δηλαδή διάβλους ώστε να περνούν τα πορίσματα των ερευνών σας γιατί η καλή σας δουλειά να αξιοποιείται και να έχει πολιτικές συνέπειες. Πώς πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αλλά ανησυχώ με πως δημιουργώ την εντύπωση ότι φτιάχνουμε εκθέσεις στις τελευταίες δύο δεκαετίες τις οποίες κανείς δεν διαβάζει και σίγουρα δεν είναι αυτή η εντύπωση που θέλω να σας αφήσω θα μπορούσα να σας δώσω και κάποια επιτυχή παραδείγματα όπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Πιστεύω ότι οι εκθέσεις επηρέασαν ας πούμε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρόκειται για ένα σχεδόν δεκαετές πρόγραμμα ε, περιβαλλοντικών πολιτικών για την Ένωση. Οπότε ε, αυτό είναι ένα πολύ θετικό ε, παράδειγμα για το οποίο θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πιστεύουμε ότι αυτό συνέβαλε στην διαρρύθμιση της πολιτικής και άμεσα και στο Συμβούλιο παρουσιάσαμε την έκθεση αυτή και στο Κοινοβούλιο, σε πολλές συνεδριάσεις μάλιστα. Υπάρχουν επιτυχίες δηλαδή όταν ε, οι αρμόδιοι μας ακούν. Μην έχετε λοιπόν την εντύπωση ότι όλα αυτά τα 20 χρόνια, όλες αυτές τις 28 εκθέσεις που σας ανέφερα κατά κάποιο τρόπο ήταν, ε, έπεσαν στο κενό. Επίσης συμμετέχουμε σε ακροάσεις ένα-δύο φορές το χρόνο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και ε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του υποβάλλει ερωτήσεις. Συμμετέχουμε σε διάφορες ειδικέ συνεδριάσεις στο Κοινοβούλιο και ναι, και εμείς, ε, ίσως θα πρέπει να αναφέρω και το εξής, και εμείς θέλουμε, όπως είπα στην αρχική μου δήλωση, να βελτιώσουμε τον αντίκτυπο των ε, εκθέσεών μας. Και εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εκπονούμε τις εκθέσεις μας ώστε να χρησιμεύουν ως βάση για την άσκηση πολιτικής. Όχι, δεν ήθελα εγώ ποτέ να υποβαθμίσω τη δουλειά σας. Ε, είναι πολύ σημαντικό Απλά θα θέλαμε και περισσότερη δουλειά ε, πιο πολύ σημασία να δίνετε στη δουλειά σας και εμείς ως πολιτικοί δεν ανταποκριθήκαμε με τον τρόπο που έπρεπε. Γι' αυτό και έγινε αυτή η Επιτροπή εδώ για να δούμε τι πήγε στραβά, τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα στον έλεγχο των εκπομπών, αλλά και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ, κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ Έχετε δεδομένα για τις εκπομπές ε, οξυδίου του αζώτου σε πραγματικές συνθήκες σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί και που κατά κατέληξε σε μία αποκλίνουσα εκτίμηση. Έχετε αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Όχι, έχουμε μια χοντρική εκτίμηση. Έχουμε κάνει κάποιες ε, χοντρικές εκτιμήσεις που δείχνουν ότι αν είχαν τηρηθεί τα όρια θα είχαν μειωθεί οι εκπομπές τουλάχιστον κατά 50%. Σε αυτή τη στιγμή, οι οδικές μεταφορές φαίνεται να είναι υπεύθυνε για το 40% του, του οξυδίου του αζότου σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό θα είχε πέσει στο 20% αν όλες οι προηγούμενες γενναίες είχαν τηρήσει τα όρια. Βέβαια, όπως σας είπα, είναι χονδρικοί υπολογισμοί. Και αυτό γιατί τα... Ε, οι διζελοκινητήρες είναι μεταγενέστεροι. Ίσως να οφείλεται και σε αυτό. Κυρία Κονέτσκα, θα ήθελα να κάνω μια περώτηση. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε πού υπήρξε το λάθος και να το διορθώσουμε. Ούτε εγώ δεν ήμουν δραστηριοποιημένη πολιτικός όταν παρουσιάσατε την πρώτη έκθεση για το, 2000, το 2005 ας πούμε. Ε, δεν υπήρξε όμως καμία αντίδραση ώστε να μπορέσουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε αυτή την έκθεση τελικά, να δούμε πώς συγκεκριμένα ε, Έπειτα από όλα, περιλημμένως αναφέρατε την εντολή, δηλαδή η βελτίωση της διαβίβασης των πληροφοριών, πώς θα θέλατε και ποιε θα είναι οι προτάσεις σας ε, ε, για να βελτιώσουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν συμφωνώ με το ότι δεν έγινε τίποτα. Θα πρέπει να δούμε αν έγινε κάτι. Γιατί διαφορετικά παραβιάζεται η καλή διαδικασία. Και έχετε κι εσεί μια ευθύνη. Γιατί όταν διαπιστώνετε ότι κάτι δεν λειτουργεί και όταν βλέπετε ότι υπάρχει απουσία ε, σεβασμού, θα έπρεπε να δούμε ε, να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ο οργανισμός περιβάλλοντος δεν συντάσσει την εντολή του. Η εντολή, του, η εντολή μας συντάσσεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο ρόλος μας είναι βασικά ε, να παρέχουμε πληροφορίες και γνώση. Αυτό το κάνουμε νομίζουμε. Εάν ε, τα ευρωπαϊκά όργανα στο μέλλον επιλέξουν να αλλάξουν την εντολή μας, Αυτό είναι θέμα των θεσμών. Επίτροπο αρμόδιο για το Περιβάλλον και οι σχετικέ δηλώσεις. Μπορώ να σας διαθέσω το έγγραφο που είπα ότι είχαμε προετοιμάσει. Σε κάποιες περιπτώσεις για να δείτε ότι όντω ε, πρόκειται για θέματα που εμεί τα έχουμε αντιμετωπίσει. Ναι, μάλιστα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας στείλετε αυτά τα έγγραφα, γιατί... Ναι, όχι, εγώ έχω μια ερώτηση στον κύριο Κράριντς. We have a law where we have a maximum speed of 50 in town. Δηλαδή, αν έχουμε ανώτατη ταχύτητα 50 μίλια, κατηγορείται το μέλος του Κοινοβουλίου αν κάποιος ε, οδηγεί με 70, εμείς έχουμε, την... Ε, έχουμε κανόνες, έχουμε νομοθεσία, έχουμε την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων επίσης που αστυνομεύει και επίσης έχουμε και 28 εθνικές υπηρεσίες που αστυνομεύουν. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα. Και θυμώνω γιατί όταν ακούμε τα στοιχεία από αυτή την υπηρεσία, 50.000 το χρόνο, 50.000 άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν. Οπότε δεν έχουμε καθόλου στοιχεία από το 2004, δηλαδή έχουμε περίπου 500.000 ανθρώπους στην Ευρώπη που σκοτώθηκαν επειδή η αστυνόμευση και η νομοθεσία που ψηφίστηκε από τα 28 κρατη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ευδοκίμησαν. Γιατί λοιπόν η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων παρά το γεγονός ότι η JRC ήδη από το 2007 είχε αποδεικτικά στοιχεία, δεν έκανε τίποτα, γιατί οι εθνικές υπηρεσίες δεν έκαναν τίποτα. Αυτό είναι το ερώτημα. Μην αποφεύγετε. Έχουμε δύο υπηρεσίες αστυνόμευσης που δεν έκαναν τίποτα. Και πάμε πίσω. Είπατε ότι έχετε ε, από το JRC ήδη συνεργασία από το 2007 το JRC ξεκίνησε να κάνει κάποιες δοκιμές οι οποίες έδειξαν ότι ε, τα αποτελέσματα ήταν πολύ, είχαν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Γιατί μεταξύ του 2007 όπου τα δεδομένα ήταν δεδομένα, ήταν διαθέσιμα και, και από την JRC και μέχρι το τέλος του 2010 όπου έγινε η πρώτη συνάντηση με τα κρατημέλη και αρχές του 2011 όπου το JRC τελικά μπόρεσε να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά του, γιατί χάσαμε τέσσερα χρόνια, 200.000 ανθρώπους δηλαδή, που σκοτώθηκαν μέσα σε, μέσα σε τέσσερα χρόνια και τίποτα δεν έγινε. Γιατί, έχετε κάποια εξήγηση. Πρέπει να ξεκινήσω μιλώντας ως υπηρεσία. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαστε εμείς σε θέση να αξιολογήσουμε την ε, αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά μία από τις παρατηρήσεις που θα κάναμε εμείς είναι ότι όταν ε, ε, μιλάμε για εποπτεία, για έλεγχο του συστήματος, εμείς συμφωνούμε με τα στοιχεία που υπευλήθησαν σε τούτη την Επιτροπή από την ICCT, όπου και λένε ότι υπάρχει κατακαιρματισμός του συστήματος ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όντως είναι διασπαρμένο, οι αρμοδιότητες είναι κατακαιρματισμένες και εντός των θεσμικών οργάνων και εντός των 28 κρατών μελών. Αλλά αυτό είναι το μοντέλο που έχει διαλέξει η Ευρώπη. Αυτό είναι η αποκεντρωμένη διακυβέρνηση. Είναι διαφορετικό από ένα σύστημα που έχουν, ας πούμε, οι ΙΠΑ, που είναι πιο κεντρικό σύστημα συμμόρφωσης και ελέγχου. Δηλαδή ο μάνατζερ της Fiat ζητάει, που ζητάει έναν ευρωπαϊκό φορέα αστυνόμευσης γιατί γιατί μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολιτικά το α, επιχείρημα αυτό λόγω διαφορών με τη Γερμανία. Αν δηλαδή η EPA μπορούσε να λειτουργήσει γρήγορα, θα το είχε κάνει. Αλλά αυτό που έχουμε είναι ότι υπήρχε και παλαιότερα 28 κατακαιρματισμένα 28 συστήματα κατακαιρματισμένα ε, μέσα στα κράτη-μέλη. Αλλά η JRC έχει τα δεδομένα ήδη από το 2007. Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων δεν τους επέτρεπε να τα δημοσιεύσουν. Ε, εσείς πώς εμπιστεύεστε ένα σύστημα όπου πάλι θα βασιστούμε σε 28 χώρες συν τον ε, υπεραστινόμο για να γίνει ο έλεγχος τελικά από την ε, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Πώς θα λειτουργήσει αυτό. Ναι, επειδή ο η πρόεδρος είπε να είμαστε και σύντομοι, ε, πρέπει να δούμε εδώ λεπτομερώ τι τις λεπτομέρειες που υπάρχουν από τι διατάξει από τον Ιανουάριο και την ε, οδηγία πλαίσιο για την έγκριση τύπου. Αυτό δεν είναι στη δική μα την εντολή, δεν είναι στη δική μα την αρμοδιότητα. Θεωρούμε ότι μπορούμε να το δούμε από απόσταση εμεί απ' έξω. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωση, Γιατί αυτό το φόρουμ ε, εφαρμογής, εκτέλεσης που συζητείται να δημιουργηθεί είναι ένα θετικό βήμα. Έχουν ε, υπάρξει και άλλες προτάσεις. Τώρα για το γενικό ερώτημά σας για την κατακαιρματισμένη ε, διοίκηση, ε, δεν είναι θέμα δικό μας για να το λύσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Εύη. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για, τον, ε, για τις διαδικασίες δοκιμών για, τις, ε, για το Άρτεμις. Στην έρση ε, σας που αναφέρετε, για, που αναφέρετε τις λεπτομέρειες για τις μεταφορές, λέτε ότι υπάρχουν και πιο ακριβείς εναλλακτικέ στον κύκλο οδήγηση για την έγκριση τύπου 4. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν στην σελίδα 25, οι, εκ, οι εκπομπές για τις διάφορες σειρές γίνονται μέσω της CADC ε, και μπορούν να, είναι πολύ διαφορετικά, πολύ πιο ψηλά τα δεδομένα από, τα τρέχοντα, από τις τρέχουσες δοκιμές για τα τζελοκίνητα οχήματα όπου οι εκπομπές ε, Euro 6 μπορεί να είναι 4,8 φορές περισσότερες από, ε, από τον ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης. Οι πληροφορίες αυτές για την καλύτερη αξιοπιστία της, ε, του κύκλου Άρτεμις, από πότε αξιολογούν τις εκπομπές ε, και από πότε είναι διαθέσιμες, μάλλον η απάντησή σας θα είναι 2004, έτσι, μήπως μπορείτε όμως να μου πείτε κάτι, γιατί μετά μπορεί να θέλω να σας θέσω και άλλη ερώτηση. Ναι, δεν είμαι σίγουρος για την ακριβή ημερομηνία, αλλά νομίζω ότι το Άρτεμις ξεκίνησε το 2006-2007, και ο λόγος για τον οποίο κάναμε αυτό το εργαστηριακό, ε, αυτή την εργαστηριακή φόρμουλα είναι για να μετράμε τις, πραγματικές, τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες. Άρα είναι πιο απαιτητικό από τον ευρωπαϊκό κύκλο με βάση τον οποίο γίνεται η έγκριση τύπου. Τώρα το πώς έγινε η όλη διαδικασία είναι ότι πιο ήταν πιο απαιτητικές οι προϋποθέσεις. Και βεβαίω δεν μα εκπλήσουν τα αποτελέσματα. Ναι, οι εκπομπέ είναι πιο ε, υψηλέ σε σχέση με τα, με τα δεδομένα που έχει μετρήσει το Artemis. Ωραία. Εσεί θεωρείτε ότι έχει υπάρξει κάποιο πρόσκομα που εμπόδισε την υιοθέτηση του Άρτεμις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κύκλο οδήγηση. Έχετε εσείς κάποια συνάντηση, κάποια επαφή, κάποια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τι ανταλλαγέ απόψεων, ναι. όχι. Δεν ε, μπλεκόμαστε εμεί σε τέτοιε συζητήσει για τον καθορισμό των κύκλων οδήγηση. Ο Άρτεμι είναι μια διαδικασία δοκιμών με βάση ερευνητικά στοιχεία. δεν είναι ε, παγκόσμιο σύστημα όπως το WLTP και το WLTC. Μπορώ να θέσω όλο ένα ερώτημα. Για τα διάφορα σενάρια που παρουσιάσατε στην εκθέσή σας, με βάση την προσωμείωση, το χειρότερο σενάριο που έχει μόνο μικρή μείωση για τους διάφορους σταθμούς ελέγχου θα, θα συμβεί με τα διζελοκίνητα γύρω ε, 6 και θα σημαίνει μόλις 30% μείωση σε σχέση με τα όρια του γύρω 5. Μπορούμε δηλαδή να υποθέσουμε ότι μέχρι το 2020 δεν θα μπορούμε να περιμένουμε να υπάρξουν μεγαλύτερες, ε, να, υπάρξουν, να υπάρξει υπέρβαση των ορίων γύρω ε, 6. Το ερώτημα σας έχει πολλές διαστάσεις. Καταρχάς, τα ε, οχήματα Euro 6 είναι καινούργια και δεν υπάρχουν και πολλά στο στόλο μας, οπότε θα χρειαστεί χρόνος για να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία. Επίσης, είναι, είναι σαφές ότι τα, ε, Euro, τα οχήματα Euro 6 έχουν ε, φτάσει τα όρια. Βρίσκονται εντό των ορίων, μάλλον. Γιατί μέχρι το 2025-2030 θα έχει υπάρξει τεράστια βελτίωση σε σχέση με του σταθμού ελέγχου για, τα, για την καταμέτρηση των εκπομπών. Βεβαίω ε, το να έχουμε καλύτερη ε, ποιότητα αέρα θα πάρει λίγο περισσότερο. Είναι ένα βήμα προς το λοιπόν. Έχουμε και τις ε, δοκιμές VRDE. Θα υπάρξουν βεβαίως και κάποιοι άλλοι παράγοντες σημαντικοί για τις ε, εκπομπές, ε, που θα, εκπομπές σε πραγματικέ συνθήκες που θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται, αλλά βεβαίω θα το παρακολουθήσουμε με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Πάμε στη δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο ε, προσκεκλημένους. Το σκάνδαλο της Volkswagen ε, μας οδήγησε σε όλη αυτή την διερεύνηση. Προς το παρόν έχουμε αυτή τη δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη, την οποία παρακολουθούμε, για διάφορους ε, κατασκευαστές όπως η Opel, η Mitsubishi, η Fiat, οι, ε, οι οποίες κατηγορούνται επίσης για παράνομη χρήση διαφόρων συστημάτων. Έχετε εσείς στοιχεία για το ποιοι είναι αυτοί οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν τέτοιες εγκαταστάσεις. Πολύ σύντομα, η απάντηση είναι όχι. Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω τότε τον κύριο Άνταμς, μήπως είναι καλύτερη η τύχη μου. Είπατε στην εισαγωγή σας ε, για τους 400.000 ε, ε, περιπτώσεις θανάτων. Μπορείτε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Ακούσαμε πολλά αριθμητικά στοιχεία εδώ, αλλά Ποιος είναι ο αντίκτυπος που έχει τελικά αυτή η τεχνολογία αν οι εκπομπές ε, ε, είναι τόσο υψηλές και αν έχουμε και τόσους θανάτους. Δηλαδή, ο αντίκτυπος 400.000 ατόμων ποιο ποσοστό αυτόν οφείλεται στις, ε, στα διζελοκίνητα οχήματα και μπορείτε να κάνετε κάποιο είδους διαφοροποίηση για το ποια είναι τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά και ποιες είναι οι, ποιος είναι ο αντίκτυπος που έχουν ε, αντιστοίχως. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. Όντως, ακούσατε πολλά αριθμητικά στοιχεία σήμερα. Για τους πρόωρους θανάτους, αυτό το 400.000 που σας είπα, έχουν να κάνουν με πρόωρους θανάτους, 70.000 θάνατοι από, ε, προεκλήθησαν από, από το διοξίδιο του αζότου. Κάτι που κάναμε τώρα για το 2015 και την έκθεση για την ποιότητα του αέρα είναι να δούμε τα ωφέλη που θα είχαμε εάν η ποιότητα του αέρα έφτανε στα όρια τα ευρωπαϊκά. Στις ε, πόλεις τώρα είμαστε πιο ψηλά. Ε, θα Μελετήσαμε το ποια θα ήταν τα ωφέλη αν φτάναμε τα ευρωπαϊκά όρια χρησιμοποίησαμε διαφορετικό σύστημα. 200.000 ε, έτη ζωής θα ήταν το όφελος σε σχέση με το κόστος. Τώρα πώς μεταφράζεται αυτό σε σχέση με τους πρόωρους θανάτους, μιλάμε για ένα περίπου 20-25% του, των 70.000 αυτών ε, πρόωρων θανάτων, μάλλον 17.000 ε, άτομα θα είχαν σωθεί αν είχαμε τα όρια τα ευρωπαϊκά σε ό,τι φορά την ποιότητα του αέρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παουλούτσι. Ε, Μάλιστα, ευχαριστώ για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Το πλαίσιο που προκύπτει επιβεβαιώνει δυστυχώς αυτό που όλοι γνώριζαν. Έχουν υπάρξει εκθέσεις, ε, ενημερώσεις και παρόλα αυτά δεν έγινε τίποτα Όλοι γνώριζαν τι ε, γινόταν και υπάρχουν και πιο λεπτομερείς ενημερώσεις για το θέμα της ευελιξίας που υπογραμμίζεται στην απάντηση στην τέταρτη ε, ερώτηση που σας υποβάλλουμε. Υπάρχουν δηλαδή ε, μεταβολές που γίνονται και αλλαγές που γίνονται εντός των εργαστηρίων. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις εκπομπές. Ευχαριστώ. <coughs> Uh, Όσον αφορά την ευελιξία, είχαμε ένα στοιχείο στον οδηγό για τις οδικές μεταφορές που παρουσιάστηκε και εδώ σε αυτή την Επιτροπή και που εξέταζε διάφορους παράγοντες και έδειχνε ότι 60% ε, του, της κατανάλωσης 16% ε, ε, μάλλον αφορούσε την κατανάλωση καυσίμου εξετάσαμε και άλλες μελέτες του ICCT για παράδειγμα και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων και μας ανησυχεί το ότι το ποσό αυτό, το ποσοστό αυτό μάλλον ε, αυξάνεται. Το 2010 ήταν 10% υψηλότερες εκπομπές, ενώ σήμερα ε, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 30-40%. Οπότε φαίνεται ότι οι κατασκευαστές ε, έχουν χρησιμοποιήσει όλο και περισσότερο αυτού του είδους ε, της ε, διατάξεις. Συγγνώμη, αλλά εγώ αναφερόμουν πιο συγκεκριμένα στη δυνατότητα να χρη... Να χρη... που χρησιμοποιείται στις δοκιμέ. Λέτε διαδικασίες τεστ σε συγκεκριμένες συνθήκε δοκιμή. Τι σημαίνει αυτό ακριβώ, σημαίνει τις ευελιξίες που χρησιμοποιούμε για να βελτιστοποιήσουμε το όχημα ανάλογα με τη δοκιμή. Ας πούμε, ε, πίεση των ελαστικών, ε, βάθος ε, των ελαστικών και διάφορα άλλα παραδείγματα ευελιξίες που θα μειωθούν μάλλον στις επόμενες δοκιμές αλλά και που συνολικά καταλήγουν σε ψηλότερες εκπομπές στον πραγματικό κόσμο. Αυτό έχουμε δει. Ευχαριστώ. Εντάξει, εντάξει. Αν τελείωσε ο χρόνος μου δεν υπάρχει πρόβλημα να σταματήσω. Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ κύριοι για τις συνεισφορές σας. Να επιστρέψω σε αυτό που είπε κάποιος από τους δύο μιλητές, δεν θυμάμαι ακριβώς, για τις μη αναμενόμενες επιπτώσεις της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών της εκ, εκπομπής αμμονίας, των οξυδίων αζότου που αυξάνονται. Από την άλλη πλευρά, η, τα τζελοκίνητα αυτοκίνητα παραμένουν πιο αποδοτικά από τα πετρελαιοκίνητα. Οπότε, ποια είναι η προτεραιότητα, γιατί μου φαίνεται ότι ε, κάνουμε κύκλους γύρω από το ίδιο ζήτημα, χωρίς να καταλήγουμε κάπου ποια θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, τι στόχο πρέπει θα πρέπει να βάλουμε για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Να ξεκινήσω λέγοντας τα επόμενα χρόνια και ο Μάρτιν να μας πει πιο βραχυπρόθεσμους μου στόχους για τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για μια διαδικασία ε, από την οποία εμείς ως οργανισμός θέλουμε να απεμπλακούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την αποδοτικότητα των ε, κινητήρων εσωτερικής καύσης και ταυτόχρονα έχουν τεθεί στόχοι για την εξάλληψη του άνθρακα από τις μεταφορές. Θα υπάρξει και σχετική πρόταση της Κομισιόν ε, το φθινόπωρο. Οπότε ο ε, δικός μας μακροπρόθεσμας στόχος είναι η πλήρης απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. Εννοείται γενικά τη μη χρήση ορυκτών καυσίμων, έτσι. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει και ο στόχος ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει να μειωθεί κατά 50% ο αριθμός των συμβατικών αυτοκινήτων και έως το 2050 δεν θα πρέπει να υπάρχουν σε αστικές περιοχές καθόλου συμβατικά αυτοκίνητα πλέον. Οπότε αυτός είναι για μας ο μακροπρόθεσμος στόχος. Η εξάλληψη του άνθρακα. Εγώ να σας πω τώρα κάποιους πιο βραχυπρόθεσμους στόχους. Το ακούσαμε και από άλλους συμμόλυτες ότι υπάρχει αυτή η, αυτή, αυτή η ισορροπία μεταξύ αερίων θερμοκηπίου, του θερμοκηπίου, ε, οξυδίων του αζότου και φαίνεται ότι δεν υπάρχει τρόπος να μειώσουμε ε, όλες τις ε, τιμές ταυτόχρονα και στον ίδιο βαθμό. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση ε, για το, επόμενο, το αμέσως επόμενο διάστημα. Κύριε Ντάνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις απαντήσεις που δώσατε μέχρι στιγμής. Θέλω να μιλήσω για τους ε, συντελεστές εκπομπών. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτούς τους συντελεστές για να εκτιμήσουν τις μειώσεις των εκπομπών. Στη σελίδα 14 όμως, ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν 300 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ε, γιοταχή αυτοκίνητα, και ο συντελεστής είναι 7, 7 αυτοκίνητα, όχι 7.000. Στην σελίδα 12 τα αποτελέσματα λέτε ότι δεν είναι και πάρα πολύ βίβαια. Μα πόσο αξιόπιστα είναι τελικά αυτά τα ευρήματα που έχετε δει. Η πρόκληση με τα νέα οχήματα και τις νέες τεχνολογίες είναι ότι όταν, με μετρήσεις και στοιχεία πραγματικών συνθήκων δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά. Εμείς ε, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλο και περισσότεροι φορείς κάνουν μετρήσεις με αυτά τα νέα οχήματα συζητιούνται εσωτερικά σε εμά οι συντελεστές αυτοί που έχουν μετρηθεί τα, το προηγούμενο διάστημα και ελπίζω μέχρι τον, το τέλος της χρονιάς να έχουμε καταλήξει σε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι τα νέα οχήματα ε, αποτελούν μια νέα πρόκληση. Ε, μήπως θα έπρεπε να, να μεγαλώσετε το δείγμα πώς είναι δυνατόν να είναι αξιόπιστες, αξιόπιστα τα στοιχεία στα οποία καταλήγεται όταν τα δείγματα είναι τόσο μικρά. Εφτά αυτοκίνητα. Ε, ο αριθμός 7 αφορά το γύρο 6, το γύρο 6. Ε, υπάρχουν πολλοί πιο ολοκληρωμένα δεδομένα για προηγούμενα πρότυπα. Ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη η επιτυχία όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, οι επιτυχίες μάλλον, ε, δεν είναι ομοιόμορφες. Υπάρχουν κάποιες κακές επιδόσεις ορισμένων νέων τύπων οχημάτων, ε, τα τα για παράδειγμα, ε, υπάρχουν διάφοροι τύποι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ανταποκριθούν στις απαιτήσει της νέας, των, των, των νέων προδιαγραφών. Ευχαριστώ. Ετέθησαν πολύ σημαντικά ερωτήματα για το γεγονός ότι εδώ και 10 χρόνια ε, προσφέρετε πληροφορίες και είπατε η ίδια, οι ίδιοι σας ότι οι πληροφορίες αυτές είναι πλέον πιο ολοκληρωμένες, χωρίς ωστόσο να ασχολείται κανείς. Το 2007 ήδη είχε συζητηθεί το θέμα των αποκλήσεων με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και με τα κράτη-μέλη. Είχαν υπάρξει καθόλου σημάδια ε, που εσείς ε, λάβατε ότι κάποιος προτίθεται να αναλάβει δράση Η βασική μας συνεργασία, που, ε, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, ε, είναι με την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, το, τη Eurostat, το Κοινό Κέντρο Έρευνας και ναι, οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος εδώ και πολλά χρόνια ήταν σαφείς ως προς τη φιλοδοξία τους να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά και όσον αφορά τις ευθύνες των κρατών μελών. Σε κάθε περίπτωση ήταν σαφής ο στόχος να αντιμετωπιστεί αυτή η απόκληση, διότι ήταν ε, γνωστό ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έθετε η οδηγία για την ποιότητα του αέρα, ήταν απαραίτητο να κλείσει αυτό το χάσμα. Ε, μάλλον η φιλοδοξία τότε δεν ήταν επαρκής. Ναι, όπως είπα σε προηγούμενη απάντησή μου, ε, έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έγινε τίποτα. Ε, ε, η δική μας εμπειρία ως οργανισμού που έχει εφαρμόσει την αρχή της πρόληψης για πολλά χρόνια είναι ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να είναι κανείς εκείνος ο οποίος επισημαίνει τα δύσκολα θέματα. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις, μελέτες περιπτώσεων ε, οι οποίες πραγματικά εκπονήθηκαν με σχετικά αργότερο ρυθμό από ό,τι θα θέλαμε, είναι αλήθεια. Οπότε για το μέλλον ε, ε, εσείς θα, θα, θα, θα υποστηρίζατε ένα ε, περιβαλλοντικό σήμα. Το ΕΚΒΑ το ξέρετε. Υπάρχει σήμανση για το διοξείδιο του άνθρακα. Φυσικά θα υποστηρίζαμε και την ιδέα να υπάρξει αντίστοιχη σήμανση για τα, για τα οξύδια του αζότου όπως και για την εθαλομίχλη. Κύριε Ζάλβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, δεν κατάλαβα. Έχω δύο ερωτήσει. Έχετε έρθει σε επαφή ω οργανισμό σε κάποια φάση τα τελευταία χρόνια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να θίξετε το θέμα των εκπομπών οξυδίου του αζότου ή για να υποδείξετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι εκπομπές οξυδίου του αζότου πολύ πάνω από τα νόμιμα όρια. I certainly in the, in the... Στο, τμήμα της ποιότητας στο αέρα οι συνάδελφοι το γνώριζαν αυτό και ήδη το 2010 έγινε σεμινάριο στην DG Περιβάλλοντος και έγινε και στη αναφορά και στην Επιτροπή ε, Ποιότητας στο αέρα εκείνο το χρόνο. Επίσης, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτική στα κρατημέλη παρακολούθησαν ε, υπό το πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ ε, παρακολούθησαν σεμινάρια και όταν τροποποιήθηκε το πρωτόκολλο εισήχθησαν και προσαρμογές ευελιξίας. Ένας από τους λόγους γι' αυτό ήταν το γεγονός ότι οι αρμόδιοι πολιτικοί γνώριζαν τις υψηλές εκπομπές οξυδίου του αζότου και, θα και ότι θα είχαν πρόβλημα στο να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους για τις εκπομπές. Ε, ευχαριστώ. Κάποιος συνάδελφος του Κοινοβουλίου εδώ ήρθε σε επαφή μαζί σας στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας για την Οδηγία 2746 για το πλαίσιο αδειοδότησης ε, αυτοκινήτων με κινητήρα, οχημάτων με κινητήρα. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν ε, για την οδηγία για τα οχήματα με κινητήρα ε, του 715 του 2007 ήρθαν σε επαφή μαζί σας, σας ρώτησαν, σας ζήτησαν επαφή, σας ζήτησαν ε, ακρόαση. Δεν γνωρίζω να υπήρξε αίτημα από κάποιον ε, βουλευτή, ευρωβουλευτή με τον οργανισμό μας, ειδικά για το θέμα της έγκριση τύπου. Δεν το γνωρίζω, γιατί δεν γνωρίζω και αν συνέβη κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αλλά δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ. Σαλτερμόζε Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να δώσετε οποιαδήποτε σύσταση για το μέλλον όσον αφορά την εξασφάλιση ότι το σύστημα εγκρίσεων τύπου θα μπορεί να εισακούσει τις ανησυχίες που εκφράζουν οι οργανισμοί, η ΜΚΟ ή οτιδήποτε. Έχετε κάποιο είδους σύσταση. Κοιτάξτε, ένα από τα ενδιαφέροντα ζητήματα είναι ε, το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και στην λήψη πολιτικών αποφάσεων. Είναι σαφέ ότι έχει υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά την αναγνώριση του προβλήματο από πλευρά των ε, αρμοδίων ε, και σίγουρα οποιαδήποτε απόφαση θα είναι ευπρόσδεξη. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η τακτική ενημέρωση των ε, ε, εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τον μέτρηση, αλλά και η κύκλη οδήγηση, όλα αυτά ανανεώνονται διαρκώς τα στοιχεία και πρέπει αυτά να παρακολουθούνται για να έχουμε πραγματικές βελτιώσεις. Εσείς λυπάστε για τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσατε πέρσι. Πιστεύετε ότι θα έχετε, πρέπει να έχετε κάνει κάτι περισσότερο για να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα περισσότερο. Όχι, ελπίζω να ήμουν σε, σε θέση να σας διαβιβάσω ένα βαθμό ταπεινοφροσύνης από πλευρά του οργανισμού μας, γιατί είπα εκεί στην εισήγησή μου ότι ε, ε, ότι ε, πήγαμε να τρέξαμε σε όλες τις εκθέσεις που αναφέρονταν σε αυτό το θέμα και σε 28 εξ αυτών ε, αναφερόταν το θέμα και το είπαμε πρόθεση να είμαι ταπεινόφρονο ότι αν μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι διαφορετικά θα θέλαμε να το γνωρίζουμε. Να ίσως για να επανέλθω και στα σχόλια κάποια μάλλον σχόλια που έγιναν νωρίτερα είναι θέμα στοχοθέτησης και διάθεσης των πληροφοριών στους ε, πολιτικούς ηθήνοντες. Αλλά και εκεί, και αναφέρομαι και στην ενημέρωση που κάναμε στις 10 Νοεμβρίου 2011 στην Επιτροπή Μεταφορών, ακόμα και τότε, δεν ξέρω πόσο πιο συγκεκριμένοι θα, θα μπορούσαμε να ήμασταν τότε. Πρόεδρος, σύντομα θέλω να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Όχι μόνο υπάρχει χάσμα μεταξύ της επιστήμης και των ηθινών των πολιτικών, αλλά υπάρχει και χάσμα ανάμεσα σε ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα. Δεν είστε ο, πρώτον, ε, ο πρώτος εκπρόσωπος επιστημονικού οργανισμού που έχουμε εδώ και όλα αυτά που ακούσαμε ήταν χρήσιμα, όμως πώς είναι δυνατόν ούτε ένας πανεπιστημιακός να μην έθεσε την ερώτηση. Εφόσον βλέπει ότι υπάρχει αυτή η διάσταση, γιατί δεν σας απασχόλησε να ζητήσετε μια εντολή από τους ανώτερους σας, ώστε να εξετάσετε το γεγονό ότι μπορεί να υπάρχει δυνατότητα συσκευών αναστολής, αφού ξέρουμε από τα τέλη του 90 ότι υπάρχουν τέτοιες συσκευές αναστολής. Αυτό είναι που μας, πραγματικά μας κάνει να μπορούμε και επανέρχονται τα ίδια ερωτήματα. Thank you, Chair. Your question is actually a question which uh, Hans Christian Andersen answered already some centuries ago. <laughs> Uh, uh, one of Ένα από τα ερωτήματα που συζητάμε εδώ. Πέραν το με κούλπα. Είναι το γιατί χάνονται πληροφορίες, γιατί δεν μαθαίνουμε αυτά που συμβαίνουν. Και Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε. Η δική σας η υπηρεσία, όταν μιλήσατε για το Διαχειριστικό Συμβούλιο με το 32 μέλη, ε, αναρωτήθηκα. 32 μέλη από 28 χώρες ε, δεν μπορεί να λειτουργεί και πολύ καλά. Οπότε ίσως να πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι και τις διάφορες δομές δεν ε, λέω ότι πρέπει να μας πείτε ότι όχι το διοικητικό μας συμβούλιο είναι χάλια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε λίγο γιατί πράγματα που συμβαίνουν δεν μαθαίνονται. Σχόλιο είναι περισσότερο, δεν είναι ερώτηση. Ναι, να απαντήσω κι εγώ με ένα σχόλιο λοιπόν. Για το Διαχειριστικό Συμβούλιο. Εμείς είμαστε μια οργάνωση που υπόκειται σε τακτές αξιολογήσεις. Η πιο πρόσφατη κατέδειξε ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα σε ό,τι αφορά των δομών είναι αρκετά υψηλή. Εδώ όμως έχω την ευκαιρία να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο για να απαντήσω και σε κάποια σχόλια που έγιναν για την εντολή μας. Ως οργάνωση, εμείς ε, θα υποστούμε και άλλη μία αξιολόγηση, την τακτική. Αξιολόγηση καλύτερης διακυβέρνησης. Οπότε ως οργάνωση η υπηρεσία περιβάλλοντος θα πρέπει να θα αξιολογηθεί για, τα, για την αποτελεσματικότητα, για την προσθέμενη αξία της, για τη συνοχή, για, την, για το κατά πόσο είναι σχετική η εντολή που έχει με τα εισαρμοδιωτές της. Ε, την καλωσορίζουμε βεβαίως αυτή την αξιολόγηση. Εμείς θέλουμε να, πάμε, να τα πάμε καλύτερα. Αλλά ίσω μέσω αυτή να μπορούμε να λύσουμε και κάποια από τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην απογευματινή συζήτηση. Η κυρία Κλού. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Το 2011 αναφορθήκατε στην έκθεση προς την Επιτροπή Μεταφορών και είπατε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία, ότι οι εκπομπές ξεπερνούν την έγκριση τύπου. Το έχετε ξαναδεί νομίζω αυτό, επαγγελμένος. Και απλώς φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ανησυχήσετε αρκετά, να θορυβηθήκατε για τα, ε, τους αριθμούς των ε, οξυδίων του αζότου που μετράτε και που είναι υψηλότερα. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό θέμα στη συζήτηση. Για τις συζητήσεις που κάνατε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή με το Κοινοβούλιο. Οι όροι παράνομοι ή ε, δεν ήταν οι συνθήκες σωστές, αναφέρθηκαν καθόλου Δηλαδή οι υποψίες σας επιβεβαιώθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Η εμπειρία που έχουμε και με τους συναδέλφους σας από την ε, Επιτροπή Μεταφορών. Δεν ξέρω αν είστε και μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Ναι, εγώ είμαι, λέει η κυρία Κλού. <laughs> Ε, πρέπει να σας πω ότι αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις που κάνουμε, ε, ετησίως υπάρχουν πολύ έντονες ε, στεναρές απόψεις στα ε, μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Εμείς ε, προσπαθήσαμε να τους ε, περάσουμε το μήνυμα της πτυχής της περιβαλλοντικής, αλλά δεν θεωρήσαμε ότι ήμασταν ο πιο καλοδεχούμενο επισκέπτης για κάποια από τα μέλη τουλάχιστον τη Επιτροπής. Μιλήσατε για, κάποια παράνομη α, δραστηριότητα. Ε, δεν μπορώ να κάνω αυτή την αξιολόγηση, αλλά δεν είχαμε καθόλου πληροφορίε ούτε στοιχεία για τις, α, ε, αυτές τις συσκευές αναστολής. Ναι, αλλά κάποιες υποψίες πρέπει να είχατε. Δεν ξέρω μήπως θεωρήσατε ότι δεν ήταν επαρκείς οι δοκιμές. Δηλαδή, κάποιος λόγος πρέπει να υπάρχει. Δεν προέκυψε από το πουθενά αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει αυξητική τάση στις ε, ε, εκπομπές. Ο νέος κύκλος ε, ευρωπαϊκό κύκλο οδήγηση ε, δεν είναι αρκετά απαιτητικό, δεν είναι αρκετά αυστηρό. Γι' αυτό επηρεάζονται οι εκπομπέ. Και θεωρείται ότι. Α, τελείωσε ο χρόνο μου, συγγνώμη. Την επόμενη φορά. Η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άργησα, με συγχωρείτε. Αλλά έρχομαι από μια εκδήλωση που είχε να κάνει με την ε, ένδια και την ποιότητα του αέρα και για τις μεταφορές μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των μεταφορών τον παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Και επίσης για τις πόλεις και τις περιφέρειες και τη σχετική πολιτική έχουμε την Ενεργειακή Ένωση. Θέλουμε να δούμε από στρατηγική πλευρά συνολικά το θέμα. Πρέπει να μελετήσουμε τι γίνεται με τις βιομηχανίες, τι γίνεται με, το, με την περιβαλλοντική πτυχή, θέλουμε να έχουμε με, μεταφορές, θέλουμε να δούμε την ποιότητα του αέρα, ε, τις εκπομπές και τις ε, επιπτώσεις στην υγεία. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει λοιπόν κοινή προσέγγιση. Είναι η, Επιτροπή, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος η καταλληλότερη να αναλάβει όλες αυτές, όλους αυτούς τους ρόλους ή θα θεωρούσατε ότι μπορεί κάποιος άλλος να κάνει την εποπτεία. Ο αέρας στην Ευρώπη σκοτώνει τους πολίτες μας. Σύμφωνα με την έκθεση για την ποιότητα του αέρα του 2015, 14.100 100 πρόοροι θάνατοι αποδόθηκαν στην έκθεση ε, σε, ε, σε διοξίδιο του αζότου μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς μπορείτε λοιπόν εσείς να ε, είσαστε ε, αποτελεσματικοί με βάση την εντολή σας ε, αν η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει δράση με βάση τα στοιχεία που έχετε εσείς. Για τα αρχικά σας σχόλια, για την ολοκληρωμένη κοινή συστημική προσέγγιση για διάφορα θέματα, φυσικά συμφωνούμε. Συνάδει αυτό που λέτε και με την έκθεση που έχουμε υποβάλει ως υπηρεσία περιβάλλοντος. Χρειάζεται διατομιακή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές ε, προκλήσεις. Τώρα, για την εντολή μας, ε, σε σχέση και με κάποιες προηγούμενε ερωτήσεις που τέθηκαν, με βάση την τρέχουσα εντολή, την οποία καθόρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δεν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε εποπτικό ρόλο, ρυθμιστικό ρόλο. Είπα πριν ότι θα, ε, στο αντικείμενο αξιολόγηση που θα ασχοληθεί ακριβώς με το θέμα της ε, εντολής μας, με την συνοχή του μέλους τομείς και όπως είπα και σε προηγούμενο ερώτημα, αν θεωρήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι πρέπει να αλλάξει η εντολή μας κάποια στιγμή στο μέλλον και πρέπει να μας δώσετε και κάποιο εποπτικό ρόλο, αυτό θα χρειαστεί πόρους, πολιτική στήριξη και να επαναλάβω κάτι που είπα πριν. Εμείς ως υπηρεσία δεν θα θέλαμε να κάνουμε να αναλάβουμε τέτοιο ρόλο εάν πρόκειται να συνδεθεί το όνομά μας με κακής ποιότητας υπηρεσίας. Ο κύριος Τούρμας. Ευχαριστώ. Να επανέλθω σε αυτό που είπατε για τις συναντήσεις ε, του 2007 με την ε, GRC. Μας υποσχεθήκατε ότι θα μας δώσετε αντίτυπα των ενημερώσεων ε, για, την, για τον κύριο Ποτότσινγκ που ήταν υπεύθυνο, ε, περιβάλλοντος τότε. Εμάς θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αν μπορούσατε να μας, έχετε, να μας δώσετε τέτοια αντίτυπα των συναντήσεών σας και με την JRC το 2004 από το 2004 μέχρι σήμερα για να καταλάβουμε πότε έγιναν δοκιμές, πότε υπήρξαν αποτελέσματα. I can just say uh, any information that we have that... Ε, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μπορώ να σας διαθέσω τα, τα έγγραφα που έχουμε. Η βιβλιογραφία που υπάρχει μπορεί να είναι διαθέσιμη και σε εσά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε πίσω στην Κοπεχάγη και θα δούμε τι στοιχεία έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τα νούμερα τώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 14.000 θανάτους, είπαμε. 50.000 πρόοροι θάνατοι μας είπατε πριν, από τη μη τήρηση των κανόνων. Αυτό είναι ετήσιο νούμερο. Είναι, δεν είναι εξωφρενικό το νούμερο αυτό. Αν δεν είναι αυτό το νούμερο εξωφρενικό, ποιο νούμερο θα ήταν. Το 50.000 προκύπτει από διάφορες πηγές. Ε, για την Ευρώπη των 28 μιλάμε. Για το 2012 είχαμε 70.000. Και ένα κομμάτι αυτών προέρχεται από τις ε, αστικές μεταφορές. Ε, παρακαλώ, μήπως μπορείτε να μας το δώσετε γραπτός και αυτό. Γιατί εδώ έχουμε νομίζω ένα σκάνδαλο τεράστιο σκάνδαλο που έχει γίνει ποτέ σε βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη και χρονολογείται από το 2004. Περιμένω λοιπόν από εσά μια χοντρική, ένα χοντρικό υπολογισμό ετήσιων πρόωρων θανάτων, γιατί είναι σημαντικό. γιατί νομίζω ότι η έκθεση σε ε, αέρα, ε, σε ε, μολυσμένο αέρα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας θανάτων. Ε, το ο αριθμός αυτός, εάν είχαν εφαρμοστεί οι κανόνες και η νομοθεσία, ποιος θα ήταν. Αυτό θέλω να μου πείτε εμένα. Μπορώ να σας στείλω κάποιους έτσι, χοντρικούς υπολογισμούς, αν θέλετε, με βάση και τα στοιχεία που έχουμε από άλλους. Ευχαριστώ. Να κλείσουμε λοιπόν, ευχαριστώντας και τον κύριο Άνταμς και τον κύριο Μακλίδη για το ανοιχτό πνεύμα που επέδειξαν για τη σύνοδο αυτή. Δεν ήταν εύκολη η ακρόαση αυτή, αλλά μας έδωσε τροφή για σκέψη και για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως προσβλέπουμε στις ευθύνε που έχει, η Σαρμοδιότητας μάλλον που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να δούμε και λίγο τα του οίκου μας. Θα υπάρξει εκτεταμένη ε, ε, έκθεση πάνω στα ευρήματα αυτά και βεβαίως αν υπάρχουν εξελίξεις με την ε, εντολή σας, ευχαριστώ να τις δούμε. Ευχαριστώ όμως που ήσασταν παρόντες, ευχαριστώ που απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας, να ρωτήσω αν έχετε κάποιο θέμα στα διάφορα να θέσετε. Δεν βλέπω να ζητά κανένα το λόγο. Σας ενημερώ λοιπόν ότι η επόμενη συνάντηση των συντονιστών θα είναι στις 19 ε, 21 ε, Ιουνίου όπου θα καθορίσουμε το πρόγραμμα του δεύτερου εξαμήνου του χρόνου. Και μετά η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής είναι στις 16 Ιουνίου. Όλη τη μέρα. Πρώτη φορά που θα έχουμε μερίσια συνάντηση.